Okay, going to Γεια σας συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορίες. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας, της κυρίας Μπρέσο, μια ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Τωρίνο από διάφορες χώρες θα μας δείτε να ψηφίζουμε. Δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουμε αρκετή ψηφοφορία. Χάσατε τη συζήτηση που έγινε το πρωί η οποία ήταν ενδιαφέρουσα νομίζω. Πρόκειται για την ψηφοφορία για το αναπτυξιακό ε, πλαίσιο μετά το 2015. Είναι σημαντική η ψηφοφορία για μας και ελπίζω να σας προκαλέσει το ενδιαφέρον. Οι καινούργιοι κανόνες του Κοινοβουλίου απαιτεί η τελική ψήφος να γίνεται ονομαστικά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, θα ήθελα να ελέγξουμε το μηχάνημα. Γιατί λόγω δύο συναδέλφων στην προηγούμενη φορά που ψηφίσαμε είχαμε δυσκολίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ό,τι θέλετε ψηφίστε. Λοιπόν, έχω 26, 27 ψηφίσαντες. Ένας επιπλέον από το ΕΛΚ αφαίρεσε τώρα την κάρτα του, οπότε είμαστε εντάξει. Πέρα της ψηφοφορίας. Δουλεύει λοιπόν το σύστημα, δεν έχουμε πρόβλημα Έχουμε ένα αριθμό συμβιβαστικών τροπολογιών. Πολλές από τις τροπολογίες καταπίπτουν λοιπόν. Θα σας ενημερώνω ε, κάθε φορά. Θα ξεκινήσουμε. Βασικά σε δύο τμήματα θα ψηφίσουμε, αν καταλαβαίνω καλά. Θα σας λέω μετά μαζί με τους αριθμούς το πρώτο τμήμα. Τώρα λοιπόν στο πρώτο τμήμα ξεκινάμε με την συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ της συμβιβαστικής 3 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 81 στη σελίδα 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 84 ε, η τελευταία στη δεύτερη σελίδα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Θα το ελέγξουμε και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. 84 για την 84 στο βάθος της σελίδας 2. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα ε, το κάνουμε για μια ακόμη φορά. Ψηφίζουμε, έχει καταπέσει 82. Ψηφίζουμε τώρα την 84 στη δεύτερη σελίδα. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 84 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε πάντες ένας επιπλέον από τους σοσιαλιστές. Λοιπόν δεκτή. 14 υπέρ 12 κατά. Περνάμε τώρα μετά από αρκετές σελίδες και πηγαίνουμε στην 7, σελίδα 7 εφόσον έχετε το ίδιο πακέτο. Λοιπόν, πρώτα περνάμε στη συμβιβαστική 4, στη σελίδα 5. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της 4. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η συμβιβαστική 4. Πηγαίνουμε στην 139. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες απερίφθη. Εκατόν σαράντα δύο. Ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 143 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 143. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 148 στη σελίδα 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Εκατόν στη σελίδα 8. Λοιπόν, 156. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 156 ψηφίζεται. 156 επαναλαμβάνω. Πέραση της ψηφοφορίας. 13 υπέρ 12 κατά Περνάμε τώρα στην 162, στην σελίδα 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 162. Ελέγχουμε, ψηφίζουμε. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή. 165 στη σελίδα 9. Ναι. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 169. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171. Υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 171. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. 153. Στην ίδια σελίδα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στο 167. Τώρα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Απερίφθη. ζητήσατε και χωρισμένη ψηφοφορία στην 190 αλλά έτσι κι αλλιώς έχει καταπέσει. Λοιπόν, πακέτο 6, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Φτάνουμε τώρα στη σελίδα 15. Α, για μια στιγμή, όχι, μια στιγμή. Πακέτο 7, πακέτο 7. Η τέταρτη στη σειρά στη σελίδα 13 διευκρινίζει πρόεδρος. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της 7. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 224. Α, όχι, έχει καταπέσει και η 224. 229. υπέρ, κατά. Νομίζω ότι δεν γίνεται δεκτή, αλλά θα ελέγξουμε. 2.29. Πέρασε τις ψηφοφορίες απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. Στη σελίδα 16 έχω την 239. Ποιοι είναι υπέρ. 239 στη σελίδα 16 του κυρίου Νίρς Ντέβα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά στην συμβιβαστική 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δύο εξήντα τέσσερα. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές δεκτή. 2.68 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.73 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 273 Τέλος. Δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική εννέα, Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε τώρα στο κάτω μέρος της σελίδας 20. Έχω την 291 υπέρ της 2.91 κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2.91 ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα. είναι το πακέτο 10, όλες οι τροπολογίες της Επιτροπής Γυναικών. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Περνάμε στο πακέτο 11, στη σελίδα 3 ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 335. Στην 335. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 335. Τέλος της ψηφοφορίας. Έχει κατα... απορριφθεί. 15 υπέρ, 12 κατά. Λοιπόν, 3.39. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 3.39. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απερίφθη. 341. Βάιρινεν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.45 Σάντσεϊ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ξαναψηφίσουμε την 345, παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, δεκτεί με μία ψήφο διαφορά. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 12. Ποιοι είναι υπέρ της 12. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τρία σαράντα πέντε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. 354, συγγνώμη, 354, για μια στιγμή, υπάρχει μια σύγχυση. Στην παράγραφο 23, 354, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, αλλά θα το ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 15 υπέρ, 13 κατά. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην 367. Λοιπόν, 367. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 367. Τέλος. 15 υπέρ 13 κατά. Περνάμε τώρα στο πακέτο 13. Ποιοι είναι υπέρ της συμβιβαστικής 13. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Την 392 τώρα. Στο βάθος της σελίδας 9 του Λουί Μισελ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 392. Πέρας ψηφοφορία ψηφοφορίας απερίφθη. Η 393. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 394 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πακέτο 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 406 στην παράγραφο 27 Γκέρεντς και Μισελ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε 406. Τέλος της ψηφοφορίας δεκτή με δύο ψήφους διαφορά. 408. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Δεκτή με μία ψήφο διαφορά. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας ΔΕΒΑ. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. 4-11. Τέλος της ψηφοφορίας για την 411 δεκτή. Πακέτο 16, ε, συμβιβαστική 16, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. Πακέτο 17, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τέσσερα πενήντα πέντε. για τις τροπολογίες Χάουταλα και Σαρτζεντίνη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στο πακέτο 2, εναλλακτική 2, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτό. Μετά περνάμε στην τροπολογία 27, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 28 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι γίνεται δεκτή αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 28 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, δεκτή. Ελέγχουμε τις τροπολογίες που έχουν ε, καταπέσει. Λοιπόν, στη σελίδα 19. Πακέτο υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Στην 16. Σλάιν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 17. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 19 τέλος δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θα ψηφίσουμε τώρα ομαδών τις αναφορές της Επιτροπής Γυναικών στο σύνολό τους. Μιλάμε για την Επιτροπή Γυναικών. Θα ψηφίσουμε on block λοιπόν όλες αυτές τις τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. δεν απορρίπτονται πραγματικά αλλά περιλαμβάνονται στις άλλες συμβιβαστικές τροπολογίες. Περνάμε τώρα στην τελική ψήφο, ονομαστική. Προσέξτε πώς θα ψηφίσετε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ και εστία. Θέλετε το λόγο μετά από το τέλος αυτής της σημαντικής ψηφοφορίας. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Νομίζω ότι πράγματι ήταν μια καλή κοινή προσπάθεια. Συνεργαστήκαμε και μείναμε στα θέματα τα οποία μας ενώνουν. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ισχυρή φωνή και στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης και τους Κιώδης για την προσπάθεια που έκαναν. αν δεν είχαμε ε, την προσπάθεια αυτή που έκαναν οι συνάδελφοι θα παιδευόμασταν μια μισή ώρα εδώ. Περνάμε τώρα. Υπάρχει άλλη μία ψηφοφορία για την διατροφή, το ψήφισμα για τη διατροφή, δεν ξέρω αν το έχετε. κοινό ψήφισμα, ψηφίσματος για τα θέματα της διατροφής της υποανάπτυξη χώρες. Θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση. Ποιοι είναι υπέρ της ερώτησης. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα περνάμε στο κείμενο της πρότασης. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Τέλος. 16 υπέρ 11 κατά. Τροπολογία 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή. 27, 26 συγγνώμη λέει πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ της 26. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 30 τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται 31. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και εδώ για την 31. Απορρίπτεται. 32. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 32 τέλος απορρίπτεται 33 ποιοι είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 33 ψηφίζουμε τέλος Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε. 34. Τέλος. Λοιπόν, απορρίπτεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Λοιπόν, για την 35 επανέρχεται η πρόεδρος. Επανερχόμεθα στην 35. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 36. All those in favor. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα την επαληθεύσουμε. 36 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεψουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 με 14. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε τη 41 Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, θα την επαληθεύσουμε. 42 άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχιτη η ψηφοφορία πέρας δεκτή 44 καταπίπτει 45 του κυρίου Ντίβα υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ το ΕΛΚ δεν κινείται κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και γίνεται δεκτή. Με άνεση. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε την ψηφοφορία πέρας δεκτή όχι καταπίπτουν. 53. Α, πρέπει να επαληθεύσουμε την ε, τροπολογία 52. 52 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. 54. Δείξτε μας υπέρ κατά. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 ντεβα υπέρ κατά θα την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 57 όχι 57 ναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά άποχες θα την επαληθεύσουμε 58 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 59 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να να παληθέψουμε. Την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Την 60, ναι. Πέρας. Απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά θα την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. 63. τρία. Τροπολογία 63 υπέρ. Κατά. Θα την επαληθεύσουμε άρχια ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές υπέρ δεκτή τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και είναι πάλι θεύμα Ναι, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 9 αρχή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας 10 υπέρ κατά. Θα την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 12. Υπέρ. Κατά. Αναποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε την 14 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 17 αρχιτή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 18 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε την 18 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 και τελευταία υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. Τροπολογία 22 άρχεται η ψηφοφορία. Α, απορρίπτεται. Τέλος πάντων τώρα. Πέρασε. Ναι, απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία για τα πρακτικά. Άρχεται η ψηφοφορία.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 leaving. I just want, I'm just going to give a minute to go so that I can give the rapporteur the floor on the next item. So you can do it in peace and quiet and not with people moving around. Περιμένουμε ένα λεπτό για να φύγει για να μιλήσει και ο εισηγητής με ησυχία. Okay, so those who are leaving, please leave quietly. We'll move. Παρακαλώ λοιπόν όσοι βγαίνουν ήρεμα. Σημείο 10, ξαναβολής από το πρωί. Α, λάθος έκανα. Με συγχωρείτε. Δικό μου λάθος. Λοιπόν, σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια. Η Επιτροπή μας βοήθησε να οριστεί το 2015 έτος της ανάπτυξης και το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ. Και η απόφαση αυτή επηρεάστηκε από την Επιτροπή μας και το σύνθημα είναι ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας, που επινοήθηκε από τα μέλη της ΔΕΒΕ. Συμπίπτει με την προθεσμία για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και θα μας δώσει την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες. Συγγνώμη, μα ε, μπορείτε να μην μιλάτε. Αν είναι να κάνετε πηγαδάκια, παρακαλώ έξω. Οπότε θα είναι μια σημαντική ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με το κοινό και οι συντονιστές μας δημιούργησαν μια μικρή ομάδα εργασίας για να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε. Έχουμε συνεδριάσει δύο φορές με τον κύριο Γκέρενς που ήταν ο Ευρωβουλευτής που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης και θα ζητήσω τον λόγο τον κύριο Γκέρενς και μετά από την Concord την πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών. Ο κύριος Γκέρενς λοιπόν έχει τον λόγο για να μας πει τις προτάσεις των συντονιστών για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστές εδώ, έτσι ώστε να προειδοποιήσει ή να ανακοινώσει το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν Ευρωπαϊκή Χρονιά Ανάπτυξης. Έχουμε σαν εταίρο μας την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θυμίζω εδώ ότι η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε και σε μια νομοθετική πράξη την οποία υπεψηφίσαμε στις αρχές του 2014. Για πρώτη φορά λοιπόν, νομίζω πρέπει να το θυμίσουμε αυτό, ...που μία πλευρά της εξωτερικής πολιτικής γίνεται αντικείμενο ε, της ευρωπαϊκής, ε, μιας ευρωπαϊκής χρονιάς. Για 12 μήνες θα έχουμε την δυνατότητα να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο την συνεργασία για την ανάπτυξη και το έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί υπογραμμίζει ακριβώς κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες θα μπορούσαμε να πάρουμε σαν Επιτροπή Ανάπτυξης στα πλαίσια της χρονιάς η οποία θα ασχοληθεί με αυτό. Σας θυμίζω επίσης ότι επιμείναμε για να δώσουμε μια κεντρική θέση στην ενότητα, στην διαδικασία που θα ακολουθήσουμε του χρόνου. Το σύνθημά μας είναι ο κόσμος μας, το μέλλον μας, η ενότητά μας. Ε, δεν τονίζουμε το κτητικό του κάθε ενός από αυτά βέβαια. Ε, εμείς προσπαθούμε να συνειδητοποιήσει ο καταναλωτής, ο οποίος φέρει την προσπάθεια της συνεργασίας και την στηρίζει, ακόμα και αν δεν είναι σωστά ενημερωμένος, λεπτομερώς ενημερωμένος. Όλες οι δημοσκοπήσεις της Eurostat και άλλα Ινστιτούτα ε, οδηγούν στο ότι η κοινή γνώμη είναι υπέρ της πολιτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Κεντρικό στόχο έχουμε την συνεκτικότητα των πολιτικών, θέμα στο οποίο έχουμε ήδη εκφραστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα της Επιτροπής μας και ορίσαμε ένα εισηγητή, πιο συγκεκριμένα μια εισηγήτρια. Τα μηνύματα κλειδιά αυτής της προεκλογικής, της εκστρατείας μάλλον, της ενημερωτικής, θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν παγκόσμιος εταίρος που έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε ένα κόσμο όλο ένα περισσότερο άλληλο εξαρτώμενο με την παγκοσμιοποίηση, με την κυκλοφορία του πλούτου και με την αύξηση δυστυχώς των ανισοτήτων. Είναι μια πρόκληση για την πολιτική ανάπτυξη και συνεργασίας, γιατί ο πολλαπλασιασμός του πλούτου δεν θα καταργήσει μόνος του την φτώχεια, χρειάζεται μια βολονταριστική πολιτική. Και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την πολιτική ανάπτυξης. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την δυνατότητα να υπογραμμίσει περαιτέρω το θέμα αυτό. Υπάρχουν αρκετοί πρωταγωνιστές και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, την εκστρατεία συγγνώμη, με ευφυή και αποτελεσματικό τρόπο. Και γι' αυτό Κάναμε πολλές συνεδριάσεις προσπαθώντας λίγο να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί μέσω συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών. Και αναφέρομαι εδώ με, τις, ε, με τους επισκέπτες προσωπικότητες πολύ γνωστές που προσκαλούνται από μέλη του Κοινοβουλίου και αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου, προσωπικότητες που έχουν μια άμεση σχέση με την πολιτική της ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν έτσι θα προσπαθήσουμε να διαχύσουμε τις ιδέες μας και η δεύτερη δυνατότητα που θα μας δοθεί είναι οι μέρες ανάπτυξης που γίνονται σε αιτήσια βάση εδώ και κάποια χρόνια στις Βρυξέλλες και εδώ θα έχουμε την δυνατότητα να οργανώσουμε ένα πάνελ υψηλού επίπεδου στα πλαίσια των ημερών ανάπτυξης. Πρέπει να επωφεληθούμε επίσης και από τις ανοιχτές θύρες στα κοινοτικά όργανα στις αρχές Μαΐου, την τη γιορτή του Αγίου Σούμαν όπως λέμε αστιαβόμενοι στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο και στις Ιλέες. Ε, παλεύουμε λοιπόν σε επίπεδο ιδεών ε, φέρνοντας στην επικαιρότητα ε, την προβληματική για την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Κάτι άλλο το οποίο περιλαμβάνεται εδώ είναι η έκθεση η Παγκόσμια Έκθεση, η Διεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015, Expo Μιλάνο 15. Έχει σαν κεντρικό στόχο την πείνα στον κόσμο και την διατροφή γενικότερα. Θα μπορούσαμε εδώ να τονίσουμε το δικαίωμα στη διατροφή. Και τέλος, έχουμε σαν εταίρος σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κοινοβούλια των κρατών μελών που έχουν και αυτά ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική μοιρασμένη αρμοδιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε επίπεδο συνεργασίας και είδαμε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν στον τομέα ας πούμε της καταπολέμησης του ιού έμπολα Υπάρχουν πολλά που μένει να ολοκληρωθούν και πρέπει να αναζητήσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Δεύτερον, έχουμε την δυνατότητα να συναντήσουμε τα κοινοβούλια των κρατών μελών και να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα, ξεκινώντας νέες μορφές συνεργασίας με τα κοινοβούλια αυτά. Εμείς να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως πρέσβεις της ανάπτυξης, να πάμε στα κοινοβούλια των κρατών μελών στις αντίστοιχες ε, ομόλογες επιτροπές τους και να κεντήσουμε θα έλεγα ένα δίκτυο δεσμών μεταξύ μας. Επιλέξαμε βέβαια τον όρο ε, πρέσβης, ακούγεται λίγο φιλόδοξο, ιδιαίτερα για τον κύριο Στήρ, ο οποίος είναι πραγματικά ένας εξαίρετος διπλωμάτης, ενώ εμείς απλά θέλουμε να προωθήσουμε την υπόθεση της ανάπτυξης και της συνεργασίας. Να μεταφέρουμε τον λόγο το καλό λοιπόν στα κοινοβούλια των κρατών μελών για τις ευκαιρίες που έχουμε να δουλέψουμε μαζί. Θα πάρουμε μέρος και σε διάφορες άλλες συναντήσεις, στην εναρκτήρια συνεδρίαση στο Αμπιτζάν τον Ιανουάριο συζητήθηκε το θέμα σήμερα και στα πλαίσια των Προέδρων. Δεν ήμουνα εδώ στη συνεδρίαση το πρωί, στους συντονιστές μάλλον. Υπάρχει και η ακρόαση για, την αηφορο, για τους στόχους της αηφορίας μία ακρόαση προβλέπεται την επόμενη άνοιξη. Euh, Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο ακρόασης στις 20 Φεβρουαρίου. Μία αντιπροσωπεία θα πρέπει να πάει επίσης στο ανατολικό τμήμα του Κονγκό, κοντά στη Ρουάντα, μία άλλη στη συνάντηση της Άντης 13 με 16 Ιουλίου. Και τέλος έχουμε και τη συνάντηση κορυφής για τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Το 2015 λοιπόν στο δεύτερο τμήμα του 15 Αυτά. Έχουμε τα, συνηθισμένα μέσα στη διάθεσή μας. Εμείς θα συναντήσουμε την επόμενη εβδομάδα εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να πετύχουμε στο στόχο μας και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για την αύξηση του επίπεδου ευαισθητοποίησης του πολίτη. Τελειώνω θυμίζοντας ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Επιτροπή μας το ότι πέτυχε να εγγράψει τη θεματολογία της ανάπτυξης ε, αυτή την εποχή η οποία είναι μια εποχή με αυξανόμενες δυσκολίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα λέγοντας ότι η αλληλεγγύη είναι εδώ, είναι αδιέρετη, έχει μια εσωτερική πλευρά και μια εξωτερική πλευρά και τα δύο πηγαίνουν μαζί. Αυτά. Αυτά. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία θα κάνουμε να μετατρέψουμε αυτή την ομοθετή πράξη σε μια πραγματική προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Μάριος Βάντες από την Concord. Πλατφόρμα που θα μας εξηγήσει τα σχετικά που είσαστε. Εκεί, πολύ καλά θα μας παρουσιάσετε ποια είναι τα σχέδια της Concord για το μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την άτυπη συνάντηση της Επιτροπής μας με την Concord. Σας ευχαριστούμε πολύ και υπάρχει δυνατότητα λοιπόν ενημέρωσης των μελών μας για αυτό το έργο. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για το καλωσόρισμα που μας απευθύνατε Σύντομα εισαγωγικά. Είμαι Ολλανδός πολίτης και εκπροσωπώ εδώ στις Βρυξέλλες σε αυτή την ακρόαση μία από τις πιο μεγάλες ανθρωπιστικές μικιο. Είμαι όμως εδώ ανάμεσά σας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Concord του ε, της πλατφόρμας αυτής των ανθρωπιστικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ευχαριστώ για την τιμή που μας προσφέρετε για να ενημερώσουμε τα μέλη για το τι συμβαίνει σε σχέση με την Concord και το τι γίνεται σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία για να εξοικονομήσουμε χρόνο, να δώσουμε μια περίληψη σε ένα σύντομο έγγραφο που ελπίζουμε ότι θα έχετε λάβει για τις διαφορετικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που σκοπεύει σε εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει η Concord και με τους εμπλεκόμενους. Έτσι λοιπόν μια συμμαχία της κοινωνίας των πολιτών για αυτές τις δράσεις. Αν θεωρείτε πρόεδρε ότι θα μπορούσε να υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και σχόλια μετά από αυτή την παρουσίαση, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα είμαι στη διάθεσή σας να σχολιάσω ή να απαντήσω. Τώρα όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη πολύ σημαντική πτυχή και είναι η περίπλοκη αντιμετώπιση της πρόκλησης του καθορισμού και του συντονισμού μιας πραγματικά ευρείας συμμαχίας συνασπισμού δράσεων από την ευρωπαϊκή κοινωνία, όχι μόνο στο επίπεδο των Βρυξελών, αλλά και στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά εμπλεκόμενοι της κοινωνίας των πολιτών ως εμπλεκόμενοι σε αυτή τη συνεργασία για την ανάπτυξη από πλευρά της, ε, ε, των Βρυξελών. Βασίζεται σε εμά σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κόνκορντ ώστε να μπορέσουμε να εμπλακούμε και να ε, εντάξουμε σε αυτή την προσπάθεια το δυνατόν περισσότερους ε, και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας και στο επίπεδο των κρατών μελών, πράγμα που κάναμε και στο παρελθόν, κάνουμε σήμερα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον. Για κάποιους τομείς της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών αυτό θα είναι εύκολο έργο, μια και είναι οργανωμένη και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο. Ο τομέας των ανθρωπιστικών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων από πλευράς ΜΚΟ, από πλευράς ανθρωπιστικής βοήθειας, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ΜΚΟ, έχουν πλατφόρμες που, λειτουργούν ήδη στο εθνικό επίπεδο και απλώνουμε το χέρι σε αυτές ώστε να συμφωνήσουμε μαζί ποιες είναι οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να γίνουν μοχλή ανάπτυξης αυτού του έργου προς τους πολίτες των κρατών τους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσουμε να τονίσουμε με τον πιο ενδεδειγμένο και σωστό τρόπο όχι μόνο τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν και τους πόρους που έχουν κατανεμηθεί για την συνεργασία, για την ανάπτυξη, αλλά και για τα αποτελέσματα που επετέχθησαν, χωρίς να αποκρύψουμε φυσικά ότι υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και είμαστε τυχεροί σε αυτό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως και με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Επιτροπή, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρώπη των Περιφερειών και σε σχέση με το έργο αυτό στα κράτη-μέλη και με τοπικές αρχές και περιφερειακές αρχές που είναι σημαντικοί εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο. Ένα πιο περίπλοκο, μια πιο περίπλοκη ομάδα εμπλεκόμενων που θέλουμε και αυτούς να φτάσουμε σε αυτούς γιατί έχουν μεγάλη σημασία να εμπλακούν είναι οι οργανώσεις που ε, καταβάλουν ήδη σήμερα προσπάθειες ώστε να μπορέσουν μέσα από τα δίκτυα αυτά να μπορέσουν να κινητοποιηθούν και να υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινότητες ε, και πυρήνες που δεν έχουν ακόμα τόσο εμπλακεί και ωστόσο ο ρόλος τους για την προαγωγή της ανάπτυξης αυτής είναι πραγματικά τεράστιος. Και μπορούμε να πούμε ότι ολόκληρα εκατομμύρια ανθρώπων ζουν στην διασπορά εκτός της ίδιας της πατρίδας τους. Η διασπορά λοιπόν αυτή έχει τεράστιο ρόλο. Έχουμε πολίτες δεύτερης και τρίτης γενεάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διασπορά. Μπορούν να είναι πηγή κεφαλαίου γνώσεων, κεφαλαίου δράσης ε, και για τις, ε, και για τις χώρες ε, προέλευσής τους και για τις χώρες υποδοχής στις οποίες ζουν. Θα ήθελα απλά να υπενθυμίσω για τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε 400 τόσα δις δολάρια που το 2013 είχαν επιμεριστεί αύξηση σε σχέση με το παρελθόν. Η επίπτωση που μπορούν να έχουν αυτά τα δίκτυα για την συνεργασία, για την ανάπτυξη δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί με κανένα τρόπο. Καμιά φορά αυτές οι οργανώσεις έχουν με τέτοιο τρόπο δράση ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν και οι κοινότητες της πατρίδας τους, αρχικής τους πατρίδας. Όμως σε σχέση με τις ΜΚΟ δεν είναι τόσο πλήρως και καλά οργανωμένες, αν είναι καν οργανωμένες και ο Henry Kissinger όταν μίλησε στη δεκαετία του 70 όταν είπε ε, σε σχέση με αυτές ε, τις ε, κοινότητες διασποράς πώς θα μπορέσουν να καθοριστούν αυτό είναι πρέπει να ενεργοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν ώστε να υποστηριχθούν οι στόχοι και η πολιτική του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε βοήθεια που προσφέρεται γι' αυτό απευθύνω έκκληση σε σχέση με τους Ευρωβουλευτές για αυτές τις δράσεις που έχετε πολίτες που ζουν στα κράτη-μέλη και αποκινούμε τα εθνικά κοινοβούλια και τα ε, κινήματα πολιτών να μας βοηθήσετε να φτάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους της διασποράς και στην ίδια σας τη χώρα ακόμα όταν υπάρχουν τέτοιες κοινότητες διασποράς. Επίσης σε σχέση με την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή σας Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το δυναμικό μας ώστε να είμαστε, να συνεχίσουμε να είμαστε υπέρμαχοι αυτών των ε, δικαιωμάτων και να υπενθυμίζουμε την ε, επιτυχή ε, έκβαση αυτών των προσπαθειών. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που θα φτάσει στους πολίτες μας και να δημιουργήσουμε αυτή την ευρύτερη μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια του έτους για την ανάπτυξη εσείς θα έχετε πολλές ευκαιρίες δημόσια να τοποθετηθείτε, να εμπλέξετε και τα εθνικά πολιτικά σας κοινοβούλια, τα πολιτικά σας κόμματα, τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα του τύπου και άλλα σημαντικά, άλλες σημαντικές ομάδες και οργανώσεις από πλευρά των χωρών σας. Ο κύριος Γκέρενς ήδη προανέφερε συγκεκριμένο αριθμό ευκαιριών που προσφέρεται για να δραστηριοποιηθούμε. Εξ ονόματος της Concord και της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ευρώπη θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής συνειδητά να χρησιμοποιείτε με συνεκτικότητα και συνέπεια αυτές τις πηγές και αυτό το δυναμικό για την ανάπτυξη, κυρίως για τους τρεις στόχους που θέλουμε να επιτευχθούν φέτος, που είναι φυσικά να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση, να αυξηθεί η γνώση των Ευρωπαίων πολιτών, όχι μόνο για το εύρος και τις διαστάσεις αυτής της προσπάθειας, αλλά και για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Να εμπλακούν οι πολίτες με κριτικό πνεύμα κριτικό πνεύμα εμπλεκόμενη σε αυτή την προσπάθεια και να προαχθεί η κοινή αλληλεγγύη, η κοινή υπεύθυνη δράση που έχουμε όλοι ως, ως καθήκον να αναλάβουμε, να διασφαλίσουμε τις, τους πόρους και την ε, άσκηση των πολιτικών μας με αλληλέγγυο τρόπο η εμβέλεια και η δυνατότητα να έχουμε αποτέλεσμα προς τους πολίτες και ε, είναι ευρύτατο το φάσμα και το εύρος αυτό για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εμείς ως εμπλεκόμενοι από την κοινωνία των πολιτών με ιδιαίτερη ε, χαρά θα σας δώσουμε στοιχεία για αυτές τις ιστορίες ε, που από τους εργαζόμενους επιτόπου μας διαβιβάζονται και μπορούν να διαχυθούν, να διαδοθούν. Έτσι θα μπορέσουν να κατανοήσουν αυτό το μήνυμα οι πολίτες της Ευρώπης με έναν εύληπτο τρόπο τρόπο, με χρήση απλής γλώσσας, γλώσσας για τους απλούς ανθρώπους μια πολύ αξιόλογη ιστορία, ένα πολύ αξιόλογο μήνυμα μπορεί να περάσει. Αυτά τα αφηγήματα τα οποία μπορούν έτσι να εμπνεύσουν και να δώσουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και να δραχθούμε των ευκαιριών χρήσης του δυναμικού μας με κοινή ευθύνη και υπευθυνότητα για έναν υγιή και δίκαιο νέο κόσμο που θέλουμε να διαμορφωθεί και να ακολουθεί ακολουθήσει στο μέλλον για τις επόμενες γενναίες. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Vanders. Um, I'm now going to give the floor to members. Um, I have... Θα δώσω το λόγο στα μέλη. Να ξεκινήσω, λέει ο κύριος Στίβ, τον συνάδελφο Γκέρντς, που με την ομάδα εργασίας του υποστήριξε τις προτάσεις αυτές δύο θέματα. Το πρώτο νομίζω ότι είναι όχι μόνο μια καλή ευκαιρία να έρθουμε κοντά στους πολίτες, αλλά να προσπαθήσουμε μαζί με τους πολίτες οι οποίοι είναι δραστήριοι στην κοινωνία των πολιτών, να φτάσουμε και αυτούς οι οποίοι ίσως στην παρούσα φάση δεν συνειδητοποιούν πλήρως τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Αν και γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών υποστηρίζουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά το σύνθημα αυτό, ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας, θα υποστηριχθεί όσο μπορούμε περισσότερο από, από ε, τους συμπολίτες μας και για τη σχέση με τα κοινοβούλια των κρατών μελών έχει μεγάλη σημασία να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Τίθεται βέβαια το θέμα του προϋπολογισμού εδώ και του σεβασμού των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με την προσπάθεια επίτευξης του στόχου το 0,7% του ΑΕΠ. Και δεύτερον, να αυξήσουμε ε, την συνειδητοποίηση του βάρους της αρχής της, ε, ε, του καθολικού συμφέροντος, του γενικού συμφέροντος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και ρόλος μας είναι να υπογραμμίσουμε αυτή τη σημαντική πλευρά. Λοιπόν, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι να ευχαριστήσω τον Σάρλ Γκερέντς και ελπίζω να πετύχει η προσπάθεια αυτή στο μέλλον. Ευχαριστώ. Χάρταλα έχει το λόγο. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Στίερ για το ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια την χρηματοδότηση και βέβαια το 0,7% δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να αναζητήσουμε νέες πηγές για χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αλλά ε, ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα για το πώς θα απευθυνθούμε στην διασπορά. Αυτό το οποίο έκανε η χώρα μου είναι πως ξεκινήσαμε ένα έργο με την ε, Διασπορά Σομαλών που υπάρχουν αναλογικά θα έλεγα αρκετοί στη χώρα μας. Συνεργαστήκαμε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και πήγαμε στην Σομαλιλάνδη Σομαλούς ε, γιατρούς ε, και νοσηλευτές ε, και υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Νορβηγία για να αντιγράψουν λίγο τον τρόπο λειτουργίας. και χρειάζονται τόσο πολλοί επαγγελματίες στις χώρες αυτές, οπότε θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να αναζητήσετε τέτοια μοντέλα. Τέλος, να πω πως νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε την δύσκολη κατάσταση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και να αναζητήσουμε τρόπους να στηρίξουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακτιβιστές που εργάζονται υπό τρομερή πίεση. Να τους ενθαρρύνουμε να, βγάλουν, να κάνουν κάποιες ομιλίες. καθώς ε, τα πράγματα αυτά δεν είναι πολύ γνωστά και συχνά αμφισβητούν ε, το νόημα του να δίνουμε λεφτά των φορολογουμένων για την πολιτική αυτή. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Έτσι και ο Σάρλς έχει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο. Ευχαριστώ Νόρμπερτ Νόιζερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Σαρλς ε, και την Αναλίτς ε, για την δουλειά που έκανε και τις ιδέες που είχε έτσι ώστε να είναι επιτυχές το 2015. Νομίζω συμφωνούμε πως το έτος αυτό το έτος δεν πρέπει να μείνει σε Στρασβούργο, Λουξεμβούργο και Βρυξέλλες αλλά στα κρατημέλη αναφέρθηκαν ήδη τα εθνικά κοινοβούλια αλλά υπάρχουν νομίζω και τοπικές ε, και περιφερειακές ε, εταιρικές σχέσεις ε, από τους Δήμους ε, στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες για το 0,7%. Σήμερα ο Bill Gates συναντάει την κυρία Μέρκελ και διέρευσε ότι η Γερμανία δεν θα φτάσει το 0,7, θα είναι γύρω στο 0,38. Και έτσι σε σύγκριση με άλλες πλούσιες χώρες ε, είναι αρκετά χαμηλά η Γερμανία. Να αναφέρω ένα καλό παράδειγμα από τη χώρα μου. Έχουμε 16 κρατήδια και έχουν βεβαίως ε, μια πολιτιστική αυτονομία, αλλά κάνουν και τα 16 κρατήδια διαγωνισμούς για το έτος ανάπτυξης. Κάτι το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε νομίζω. Τέλος, είπαμε πως χρειαζόμαστε προώθηση. Εάν τα καταφέρουμε λοιπόν ε, σε 15 μέρες ο Πάπας Φραγκίσκος ε, στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να πει πως είναι ένα ιδιαίτερο έτος το έτος αυτό για την Ευρώπη θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι την ομιλία της ε, Λαμπεδούζας. Ε, εγώ ξέρω βεβαίως πως οι υπηρεσίες πρωτοκόλλου του Μάρτιν Σούλτς και του Βατικανού είναι σε επαφή Οπότε πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ομιλία του Πάπα. Και εάν αναφέρει νομίζω το ευρωπαϊκό αυτό έτος θα έχουμε κάνει μια καλή δουλειά και μια καλή αρχή για το 2015. Ευχαριστώ Νέτς Ντίβα. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο για να ξέρω. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον Charles Gerens θα ήθελα να συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και πλαισίωσε έτσι το έργο της Επιτροπής μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στην Επιτροπή μας εδώ είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα θα έλεγα. Γιατί όλοι είμαστε υπέρ αυτών των καλών πραγμάτων να βοηθάμε τους αναξιοπαθούντες ε, ανεξαρτήτως των πολιτικών μας απόψεων. Γιατί έχουμε κάποιες κοινέ αξίες για τις αναψώμενες χώρες. Αλλά αν δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά τη χώρα μου, αυτή τη στιγμή είμαστε, είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Και είναι εκπληκτικό το ότι η Επιτροπή μας ε, δεν έχει αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι. Για τον κύριο Κάμερον αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπει θετικά και εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε το 0,7% για να δώσουμε ακριβώ τη βοήθεια και να βοηθήσουμε τις ανθρώπινες χώρες. Αν δούμε μόλις ε, άλλες περιοχές της Ένωσης, που δεν έχουν σχέση με το θέμα αυτό, ε, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. την Για την Ουκρανία δεν συμφωνούμε, είναι εξωτερική πολιτική τίποτα, διαφορετικές απόψεις, ε, καμία ενότητα. Δια πολλές διαφωνίες, αλλά ο μόνος τομέας στον οποίον όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συμφωνούν είναι ακριβώς η ανάπτυξη. Είμαστε, υπ' αυτή την έννοια, μια τεράστια μικιό. Είμαστε ικανοποιημένοι εμείς τα κράτη-μέλη όλοι. Γιατί λοιπόν δεν το εκμεταλλευόμαστε. Γιατί δεν ακουγόμαστε. Κύριος είδε. Είμαστε σημαντική επιτροπή, κάνουμε ένα θετικό έργο και μας θεωρούν εδώ πέρα μια ομάδα έτσι λίγο περίεργων που κάνουν τα δικά τους εκεί στη γωνία ενώ οι σημαντικοί άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα εδώ. Και όταν μιλάμε για το συμφέρον των κρατών μελών δεν σημαίνει τίποτα τελικά. Είμαι σίγουρος πως η ΑΦΕΤ ε, ασχολείται με την Ουκρανία, αλλά κάθε κράτο μέλος διαφωνεί. Για τη Ρωσία το ίδιο, για το Ιράν το ίδιο. Και τα πυρηνικά και το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Αλλά όταν μιλάμε για την ανάπτυξη. Ε, είμαστε ενωμένοι. Εμείς πρέπει να κάνουμε κουμάντο θεωρώ εγώ. Σοβαρά μιλάω. Νομίζω πως... Ε, είναι η πιο εστιασμένη και οργανωμένη προσπάθεια εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν ο Τσάρλς να σκεφτεί όχι το 2015 αλλά πέρα από το 2015. Αν δηλαδή είναι να λέμε ότι κάνει κάτι καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το, αυτό κάνει. Και εγώ είμαι και ευρωσκεπτικιστής, έτσι. Ευχαριστούμε. Ναι, θα τα πούμε στις άλλες επιτροπές ότι πλέον έχουμε στόχο να κυβερνήσουμε ολόκληρη την Ένωση. Λοιπόν, κύριος Γιάντσεν. Ναι. Πράγματι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ανθρώπους που συνεργάστηκαν για το έτος αυτό αναπτυξιακής συνεργασίας γιατί νομίζω πως ε, λίγες ε, δραστηριότητες ε, συνεισφέρουν στην στον ευρωσκεπτικισμό σου αυτό το θέμα τεχνητό ενδιαφέρον που πρέπει να δημιουργηθεί για τεχνητά ζητήματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χώρες ε, που πρέπει να συνεισφέρουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε όλο και περισσότερο και νομίζω πως ε, είναι ένα δώρο Θεού ε, το έτος αυτό ε, ανάπτυξης για τους ε, ευρωσκεπτικιστές. Επίσης, όταν μιλάτε για οργανισμού, οργανώσεις της διασποράς, ε, δεν νομίζω πως αυτός ο οποίος σκέφτηκε αυτόν τον όρο έχει ιδέα του τι γίνεται σε αυτές τις οργανώσεις αυτή τη στιγμή και ελπίζω να παραμείνει έτσι αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Um, thank um, Ευχαριστώ. Προτού δώσω τον λόγο σε άλλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να τοποθετηθεί. Εσείς παρακαλώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σύντομη ενημέρωση, επικαιροποίηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς και όπως αναφέρθηκε, πολύ κοντά βρισκόμαστε στην ε, επικαιροποίηση και ανανέωση αυτού του έργου. Με ικανοποιητικό τρόπο το βλέπουμε αυτό και είναι και μια κοινή προσπάθεια, μια κοινή πρόκληση και γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό. Σύντομα θέλω να πω ότι εργαστήκαμε εμεί από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσουμε ότι από πλευράς επικοινωνία με όλων αυτών και εκεί επικεντρώνομαι θα δράσουμε από την 1η Ιανουαρίου ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί ε, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θέλουν και οι, πο, πολιτικής που θα ακολουθηθούν να ενταχθούν και είναι αυτό κάτι το οποίο έχει και τον λόγο του και εργάζονται σκληρά οι, τα στελέχη από τη Γενική Διεύθυνση ώστε να ενταχθούν και αυτές οι πτυχές από του χρόνου. Θα είναι ειδικό έτος το 2015 για όλους εμάς για διαφορετικούς και πολλούς λόγους, πολυσχηδείς λόγους. Είναι μια ευκαιρία για μας ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεκτική, συνεπή πολιτική για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Και είναι μια, ένας τρόπος να ευαισθητοποιήσουμε και άλλους και να φτάσουμε σε εκείνους που ε, έχουν στραφεί προς την συνεργασία για την ανάπτυξη. Έχουμε ο κόσμος, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας ως σύνθημα το λάβαμε ιδιαίτερα υπόψη στο σχεδιασμό του τι θα κάναμε σε σχέση με αυτά τα έργα, αυτούς τους στόχους, στην επικοινωνία μας, μια και είναι ένας αλληλεξαρτώμενος κόσμος και εργαζόμενοι επί των κυριότερων στοιχείων της εκστρατείας που θα ξεκινήσει δόθηκε και η ιδέα πριν από 1,5 χρόνο και σε σχέση με τον κύριο Γκέρετς όταν συζητούσαμε στο γραφείο του πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε εκείνους τους πολίτες που ε, δεν ενδιαφέρονται ήδη και δεν έχουν εξοικειωθεί με αριθμούς, μεγέθη κτλ. Και από τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ε, και ευαισθητοποίησης ε, θα μπορέσουμε να δράσουμε. Είναι λοιπόν μια κοινή προσπάθεια που θα πρέπει να μεταφράζεται και στα μέσα και εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιούμε την ιστοσελίδα, το διαδίκτυο, τις ε, πύλες, ε, τις διαδικτυακές. Ε, θα επικεντρωθούμε υπογραμμίζοντας αυτό το ότι δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες που συμμετέχουν, αλλά θα πρέπει να θεωρείται κτήμα και ιδιοκτησία όλων που ενδιαφέρονται στη συνεργασία για την ανάπτυξη και όχι μόνο της Επιτροπής της Βρυξέλλες. Συνεργαστήκαμε και με τους εθνικούς συντονιστές των κρατών μελών. Έχουμε από 27 κράτη-μέλη εθνικά προγράμματα συντονιστικά και δράσεις. Συμπεριλαμβάνονται λοιπόν και υπάρχει εδώ ο δεσμός, η δυνατότητα ε, διαμεσολάβησης και συνεργασίας με τα κρατη και εμπλοκή, μας, εμπλοκή τους ε, από όλα τα κρατη και την εργαλειοθήκη που αναπτύξαμε ευχαρίστως μπορούμε να σας την διαθέσουμε ένα ε, ζωντανό εργαλείο, αποτελεσματικό εργαλείο για να μπορέσουμε να δούμε τι θα μπορέσει να γίνει στα κράτη-μέλη. Θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η προσπάθεια ώστε η συνεργασία για την ανάπτυξη να φτάσει στα νοικοκυριά, στα σπίτια, στο ίδιο το σαλόνι του κάθε σπιτιού ώστε κάθε οικογένεια, κάθε νοικοκυριό να ευαισθητοποιηθεί να διασφαλίσουμε έτσι ότι θα βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο δράσης και θα μπορούμε να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε αποτελεσματικά. Δίνοντας όμως ταυτόχρονα την δυνατότητα με φάνταστο δημιουργικό τρόπο η δημιουργικότητα των πολιτών να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια δημιουργικά και αποτελεσματικά να φτάσουμε στο δυνατόν περισσότερους πολίτες. Ευχαριστώ. ευχαριστώ να πούμε στους συναδέλφους ότι Ελπίζουμε ότι αυτή η εργαλειοθήκη που είπατε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ευρωβουλευτές θα έχουμε μια συνάντηση και σε σχέση με την ε, δυνατότητα επικοινωνίας, σε σχέση με τα κονδύλια που θα μπορούν να ε, διατεθούν και δυνατότητες που θα μπορούν να διατεθούν εργαλειοθήκες από κρατών μελών θα πρέπει να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες και να συντονιστούμε για το πώς θα λειτουργήσουν αυτά. Ο κύριος Γκέρενς τώρα παρακαλώ θα έχει τον λόγο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ξέχασα πιο πριν, Πρόεδρε, στην εισαγωγή μου την εισαγωγή, στην εισαγωγή μου την συνεισφορά αυτών των ανθρώπων να την αναφέρω που είναι πολύ σημαντική για αυτές τις πρωτοβουλίες που από την Κονκόρδια μπορούν να υποστηριχθούν. Ευχαριστώ λοιπόν για το ότι από πλευράς της ε, της Κονκόρδια υπάρχει αυτός ο πυλώνας ώστε για το 2015 να δράσουμε αποτελεσματικά. Ο συνάδελφος έχει δίκιο όταν είπε ότι είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να πισθούν και με εφάνταστο δημιουργικό τρόπο να δράσουμε. Ο εφάνταστος δημιουργικός τρόπος που μπορεί να μας εμπνεύσει πολυσχηδός ώστε αυτά να ενταχθούν αποτελεσματικά. Η κυρία Χάουταλα τόνισε ότι το 0,7% του ΑΕΠ πρέπει να μπορέσει να επιτευχθεί και να το υπερβούμε. Νέες πηγές χρηματοδότησης είναι σημαντικό να διασφαλιστούν. Και τόνισε η κυρία αλλά επίσης το δυναμικό της διασποράς στις διαφορετικές χώρες, ώστε να ανοίξουν περισσότεροι ορίζοντες και δυνατότητες και να διασυνδεθούμε μεταξύ μας. Είμαι πρόθυμος να υποστηρίξω αυτή την πρωτοβουλία και αυτή τη δυνατότητα

και από πλευράς άλλου Ευρωβουλευτού αναφέρθηκε ότι φυσικά τα κράτη-μέλη πόρο απέχουν ακόμα από το να πετύχουν όλα όσα απαιτούνται ιδιαίτερα σε σχέση με το αναγκαίο ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ που θα χορηγείται στην συνεργασία την ανάπτυξη. Και ο Άγιος Πατήρ, ο Ποντίφικας, ο Πάπας Φραγκίσκος μπορεί ίσως να συνεισφέρει, να πείσει εκείνους που δεν πίστηκαν ακόμα να προσυπογράψουν αυτό το έγγραφο και συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη είπαν ότι είναι σημαντικό κάτι που ανήκει στα κεκτημένα, τα επιτεύγματα, μεγάλα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον βρέθηκαν και τα σωστά λόγια με τα οποία εξέφρασε αυτό. Είπε ότι σε αυτή την πολιτική πρόκειται για μια συνενετική προσπάθεια και αν συγκρίνει κανείς άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκρίνοντας με την εξωτερική πολιτική έχει δίκιο. Γιατί να μην είμαστε πιο φιλόδοξοι ιδιαίτερα όσον αφορά τα διεθνή φόρα και τους διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσάς Γιάνσεν για την παρέμβασή σας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και από πλευράς Κονκόρντ γιατί εργαστήκατε όλοι αποτελεσματικά καταβάλατε προσπάθειες με κάθε τρόπο ώστε αυτή η πρωτοβουλία να υποστηριχθεί και να ενδυναμωθεί αναφέρθηκε ότι οι ιστορίες αυτές, τα αφηγήματα αυτά πρέπει να είναι χρήσιμα για να περάσει το μήνυμα που θέλουμε να περάσει. Συμφωνούμε με αυτή την τοποθέτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μια εκδήλωση τον Ιούλιο νομίζω ήταν, μας είχε προσκαλέσει, επρόκειτο ιδιαίτερα για έναν ghostwriter, για έναν δηλαδή συντάκτη λόγων ε, από πλευράς ε, του πολιτικού προϊσταμένου του που συντάσσει τέτοιου είδους ε, λόγους. Είναι σημαντικό λοιπόν το αφήγημα, το αφήγημα που πρέπει να μπορέσει να διαδοθεί και να περάσει το μήνυμα και στις συναντήσεις ε, συντονιστών και συναντήσεις με πρέσβεις υπήρχαν δυνατότητες, οι, άλλοι, οι μεν ήταν υπέρ, οι άλλοι όχι τόσο πολύ. Ωστόσο υπήρχε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα επιχείρημα το οποίο παρουσιάστηκε ότι σε σχέση με αυτή την παρουσίαση ε, και τοποθέτηση από πλευράς ενός πρέσβη, ενός Γάλλου πρέσβη αναφέρθηκε είχε τη συνήθεια να πει ότι ο προηγούμενος μου ήταν παλιάνθρωπος, ε, ο διάδοχός μου πρέπει όμως ε, να μπορέσει να ε, συνεχίσει με καλύτερο τρόπο μετά από μένα. Πρόκειται λοιπόν για ένα αφήγημα στο οποίο θέλουμε να εντάξουμε με τον πιο θετικό τρόπο ένα σημαντικό θεματολογικό ζήτημα θεματολογία που θα μας απασχολήσει το επόμενο έτος 2015 διαρκέστερα. Θέλω να εκφράσω μια επιθυμία και να ολοκληρώσω με αυτήν το πιο ουσιώδες νομίζω. Το 2015 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Γι' αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι μας να υπάρχουν διαρθρωτικές βελτιώσεις, επαρκείς βελτιώσεις που θα επιτευχθούν ώστε να μπορέσουμε με αυτό αυτήν την προσέγγιση να έχουμε μια πιο θετική δράση και για τα επόμενα έτη μελλοντικά, για το απότερο μέλλον, μια πολιτική που θα εδράζεται στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πνεύμα και στην καρδιά των πολιτών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 Madame la Présidente. Euh, les rapports sur les travaux ACP... ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Οι εκθέσεις αυτές έχουν ε, πλέον γίνει συνηθισμένες. Αυτή βέβαια είναι λίγο ξεχωριστή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, α, η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ΑΚΕ περνάει μέσα από μια συνειδιοκτησία θα έλεγα και των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το οποίο από ό,τι νομίζω δεν ελέγχεται ιδιαίτερα από τα κοινοβουλευτικά όργανα. Και όταν μιλάω για κοινοβουλευτικά όργανα ε, πρέπει να υπάρχουν περίπου 100 τέτοια που θα έπρεπε να ελέγχουν το ταμείο αυτό τα κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ από τη μία, διότι εμπλέκονται, είπαμε είναι συνειδιοκτήτες, είναι η μία εμπλεκόμενη πλευρά και από την άλλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών. Τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης είναι κάτι το οποίο ελέγχεται όχι από αυτά αλλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα από τη συνθήκη να το κάνει, γιατί παραμένει όπως είπαμε σύν η ιδιοκτησία των κρατών μελών. Υπάρχει εδώ ένα επίπεδο έλλειψης οργάνωσης σε υψηλό βαθμό, κάτι το οποίο που εμποδίζει τη λειτουργία τη σωστή του δημοκρατικού ελέγχου, του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το λέγω αυτό εισαγωγικά για να κατανοήσετε ότι δεν απαγορεύεται βέβαια σε ένα κοινοβούλιο να ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες ή να δώσει μια κάποια όθηση. Αυτό κάνει και η μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση. Τίποτα δεν μας εμποδίζει εμάς να θέτουμε κάποια ερωτηματικά παρότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα τον προϋπολογισμό τους Μπορούμε παρόλα αυτά να συνεισφέρουμε κάποιες φωνές κριτικής, λογικής στα πλαίσια της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Θα ξεκινήσω με ένα νέο καλό, ότι υπήρξαν δύο αντιδράσεις στην έκθεσή μου, η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών είναι η επόμενη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα από τώρα, Υπάρχουν όμως δύο συνάδελφοι οι οποίοι διάβασαν την έκθεση. Αυτό είναι καλό νέο. Ε, και αν σκεφτεί κανείς ότι και οι βοηθοί τους το διάβασαν, αυτό σημαίνει ότι ήδη τέσσερις ξέρουν τι γράφω. Και είμαι θετικός άνθρωπος και ξεκινώ με την ιδέα ότι αυτοί που δεν διάβασαν την έκθεση και που δεν κατέθεσαν τροπολογίες, ίσως και κάτι να διάβασαν και να τη βρήκαν εξαιρετική. Αυτά για τα θετικά. Τώρα, τα αρνητικά. Το κακό είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την διοργάνωση των συνεδριάσεών μας. Ένα κράτος μέλος δεν ήταν σε θέση να οργανώσει, είπε το ευρωπαϊκό κομμάτι, των ΑΚΕ, εδώ και λίγα χρόνια. Κάποια άλλα κράτη έχουν την τάση να κάνουν το ίδιο και αυτά. έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι αυτός που θα οργανώσει τις διασκέψεις αυτές. Έχουμε λοιπόν συνηθίσει με αφορμή αυτές τις συναντήσεις να οργανώνουμε την συνέλευση στην χώρα η οποία συμπίπτει με την Προεδρία του Συμβουλίου έτσι ώστε η χώρα αυτή να έρχεται κοντά στην προβληματική των χωρών ΑΚΕ. Στο μέλλον όμως από ό,τι φαίνεται οι περισσότερες συνεδριάσεις θα γίνονται στις Βρυξέλλες και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την σωστή ενημέρωση των πολιτών. Και είναι και κάτι το οποίο βρίσκω ότι είναι αντίθετο με αυτά τα οποία είχαμε πει παλιότερα για την αυξημένη συνειδητοποίηση των πολιτών στα θέματα της ανάπτυξης. Υπάρχει επίσης και κάτι το επιπλέον που πρέπει να πούμε εδώ. Η έκθεση αυτή καλύπτει ένα χρόνο. Εδώ καλύπτει και το 12 και το 13. Δεν είναι κάτι το τρομερό βέβαια. Σημασία έχει ότι το θέμα καλύπτεται μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επιμένουμε στο ψήφισμα στην μεγαλύτερη εμπλοκή των συμπροέδρων ε, στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου Υπουργών. Όπως συμβαίνει και στα ευρωπαϊκά όργανα, το Συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάρει το λόγο και να πάρει μέρος σε ένα τμήμα των εργασιών και γι' αυτό θα θέλαμε και οι συμπρόεδροι να έχουν την δυνατότητα να είναι παρόντες ε, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου να πάρουν το λόγο. Νομίζω ότι αυτά έχω να πω στα πλαίσια της συγκεκριμένη έκθεσης. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κάτι. Εσείς να μου το θυμίσετε αν κάτι έχω ξεχάσει. Εάν κάτι παρέλειψα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ευχαριστώντας τον κύριο Πόγκα και τον κύριο Μισελ που ήδη κατέθεσαν τις τροπολογίες τους ελπίζοντας ότι όπως είπα και άλλοι διάβασαν την έκθεση και μπορεί και να αντιδράσουν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πράγματι περισσότεροι διαβάζουν την έκθεση πριν από την κατάθεση των τροπολογιών. Πόγκα, Μάνσκου και Ντίβα έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Πόγκα είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρεντς για την εξαιρετική δουλειά που έκανε για τις εργασίες ε, γύρω από την μεικτή κοινοβουλευτική παρουσιάζει με σωστό τρόπο τις εργασίες της ε, ισομερούς λοιπόν για τα έτη 2012 και 2013. Όπως λέγεται στην έκθεση, ε, τα και είναι πραγματικά ένας χώρος πολιτικού διαλόγου βορρά και νότου. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις εργασίες αυτές. Λοιπόν, κατέθεσα ορισμένες τροπολογίες για να υπενθυμίσω στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να επικυρώσουν τη συμφωνία του Κοτονού, την αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού και να ζητήσω την αλλαγή της απόφασης του Προεδρείου του Κοινοβουλίου έτσι ώστε οι συνεργάτες μας να μπορούν να μας ενισχύουν κατά τη διάρκεια των Ολομελιών. Είναι μια απόφαση που είχε ληφθεί πέρυσι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι συνεργάτες μας δεν μπορούν πλέον να μας συνοδεύουν στους τόπους εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παρμόσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω και εγώ στον κύριο Γκέρντς ότι διάβασα με πολύ προσοχή την έκθεσή σας και αν κάποιος ένας και μόνος το διάβαζε εγώ θα ήμουν, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ήδη δύο. Η έκθεση αυτή είναι μια εξαιρετική βάση εργασίας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρεια στην παρούσα φάση. Και στην, στο ψήφισμα το οποίο είχε έχει, στα ψηφίσματα τα οποία έχει υιοθετήσει η μεικτή κοινοβουλευτική τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία με προκάλεσαν θα έλεγα. Θα συμφωνώ να πω ότι έχετε δίκιο υπογραμμίζοντας το αρνητικό φαινόμενο και προηγούμενο της Ιρλανδίας και της Ελλάδας που δεν οργανώνουν στο έδαφος τους, δεν οργάνωσαν στο έδαφος τους όταν ήταν πρόεδροι του Συμβουλίου ε, θεωρούμε ότι είναι κάτι τέτοιο λυπηρό και είναι σαφές ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος του Συμβουλίου απέναντι στις, στις χώρες ΑΚΕ και στα όργανα ΑΚΕ είναι κάτι το αρνητικό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε σαν πολύ σημαντικό. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας πρέπει να τύχουν περισσότερης προσοχής. Εξάλλου, για να μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο τις εργασίες των ΑΚΕ. Συμφωνούμε μαζί τους λέγοντας ότι οι συμπρόεδροι θα πρέπει να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Μικτού Συμβουλίου ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στις εργασίες του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι σοσιαλιστές θα ήθελαν να κάνουν λοιπόν κάποιες προτάσεις για να βελτιώσουν αυτήν την έκθεση και θα λάβετε κάποιες τροπολογίες από πλευράς μας. Πρώτον, τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας στα πλαίσια του JPC με στόχο να εργαστεί για το μέλλον της εταιρικής σχέσης μετά το 2020. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι κρίσιμα στον καθορισμό του μέλλοντος των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες ΑΚΕ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, η μεικτή κοινοβουλευτική πρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει στην πορεία αυτή. Δεύτερον, στην προσπάθεια ενίσχυσης ε, της ε, νομιμοποίησης, της διαδικασίας νομιμοποίησης του JPC πρέπει να οριστούν δύο μόνιμοι εισηγητές για την συμβατότητα των πολιτικών για την ανάπτυξη. Ο ρόλος τους θα είναι να διασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή του άρθρου 12 της Συμφωνίας του Κοτονού που αναθεωρήθηκε το 2010. Τελειώνοντας, θα ήταν ενδιαφέρον οι εισηγητές να αναφερθούν στα όρια της χρήσης του παραγράφου 4 του άρθρου 16 του κανονισμού JPC. Αναφέρομαι εδώ στην διαδικασία ψηφοφορίας που μερικές φορές μπλοκάρει τις πρωτοβουλίες. Λοιπόν αυτές είναι οι παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Θα καταθέσω γραπτές προτάσεις ε, εξ ονόματος ε, του συνεισηγητή της ομάδας μου. Ευχαριστώ Νέα Στίβα και μετά Νόιζερ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέρνης για την έκθεσή σας. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι το εξής. Εμείς το λέμε ε, το μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση και 30 τόσα χρόνια. Εγώ πάντα είχα την εντύπωση πως το πρώτο καθήκον ενός κοινοβουλίου είναι να ελέγχει τον προπολογισμό. Εδώ πέρα όμως έχουμε κάτι το μοναδικό. Είναι η μοναδική κοινοβουλευτική συνέλευση που δεν έχει προπολογισμό να ελέγξει. αλλιώ τι κάνουμε, δηλαδή εδώ. Καφενείο είμαστε. Ερχόμαστε και μιλάμε. Υπάρχει προπολογισμό που δεν ελέγχει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι προπολογισμό της Κομισιόν, ο οποίος ελέγχεται αρκετά από το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και δεν ελέγχεται. Υποτίθεται τον ελέγχουν τα κοινοβούλια των κρατών μελών, δεν είναι μικρό ποσά. 23 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια. Αν δείτε όμως το ότι γίνεται στα κοινοβουλία των κρατών μελών και στη Βουλή των Κοινοτήτων, δεν ασχολούνται πάρα πολύ. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά που τα δίνουμε στην Κομισιόν να τα ξοδέψει και δεν τα ελέγχει κανείς. Και υπάρχει μια κοινοβουλευτική διάσκεψη που βολτάρει ανά την Ιφίλιο ή τέλο πάντων αυτό έκανε 100.000 ευρώ για τις συνεδριάσεις και δεν μπορεί να ελέγξει τον προπολογισμό. Προφανώς ε, οι δαπάνες ε, που κάνει η Κομισιόν πρέπει τουλάχιστον να υπόκεινται σε έλεγχο ακόμα και αν δεν μπορούμε να πούμε πού θα δαπανηθούν τα λεφτά γιατί αυτό είναι δουλειά των ε, κοινοβουλίων των κρατών μελών δεν ζητάμε να αρχίσουμε να μοιράζουμε τα λεφτά, γιατί για να τα μοιράζουμε πρέπει να τα δίνουμε όλα και δεν τα δίνουν οι χώρε ΑΚΕ. Οπότε η κατανομή είναι άλλο θέμα. αλλά τουλάχιστον να ελέγχουμε που πάνε. Τσαρλ! Ευχαριστώ κύριε Ντέβα. Στις νέες ομάδες εργασίας το Κοινοβούλιο εξετάζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Συμφωνώ μαζί σας όμως πως μπορούμε να μιλήσουμε με το Προεδρείο της ΑΚΕ πριν από 7 χρόνια το κοιτάγαμε αυτό μαζί με τους συναδέλφους από τις χώρες ΑΚΕ. Ε, μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως λίγο περισσότερο. Νόρμπερτ Νόιζερ και μετά Ενρίκη Γκερέρο. Από εμένα και από εμένα να ευχαριστώ στον Τσάρλς Κέρνς. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε πολλά, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο ο Τσάρλς Κέρνς τα λέει στα ράτα και το βλέπουμε και σε αυτή την έκθεση. Και βεβαίως μετά την κοινή συνέλευση και τις εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών να υπενθυμίσω πως επί Ιρλανδικής Προεδρίας για πρώτη φορά μια χώρα αρνήθηκε να φιλοξενήσει τη διάσκεψη. Κάτι το οποίο θα κόστιζε λίγα πράγματα στην Ιρλανδία, αλλά θα τις ε, προσέδιδε διεθνές κύρος. Και το ίδιο έκανε και η Ελλάδα μετά. Αυτό αναφέρεται στο σημείο 2 και νομίζω πως πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μην συνεχίσουν αυτή την πρακτική. Το 2014 και οι δύο συνεδριάσεις ήταν στην Ευρώπη. Η πρώτη ήταν την άνοιξη στο Στρασβούργο, η δεύτερη θα γίνει τώρα τέλη Νοεμβρίου πάλι στο Στρασβούργο. Και η κοινή συνέλευση, το Προεδρείο αποφάσισε του χρόνου και οι δύο να μην γίνουν στην Ευρώπη, οι δύο συναντήσεις, αλλά στις χώρες ΑΚΕ οι χώρες ακεσκίζονται για να φιλοξενήσουν την ε, συνεδρίαση. Γιατί θεωρούν πως κερδίζουν με το να φιλοξενήσουν αυτή τη διεθνή διάσκεψη και εμείς οι Ευρωπαίοι έτσι είμαστε πολύ χαλαροί. Οπότε έχουμε πάλι ένα χρόνο στη διάθεσή μας για να ασκήσουμε λίγη πίεση στα κράτη-μέλη. Τελευταίο σημείο. Πρέπει ως βουλευτές και εμείς ε, να κάνουμε κάτι. Δεν συμμετέχουν πολλοί οι συνάδελφοι, ειδικά αν έχουμε συνεδριάσει επιτροπών στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και εδώ πέρα πρέπει κάτι να γίνει για να παραμείνουμε και αξιόπιστοι. Ευχαριστώ και Γκερέρο τελευταίος. Σε ευχαριστώ ο λόγος για τον οποίο πολλοί ευρωβουλευτές και εγώ ίδιος κάποια στιγμή διαβάζουμε αυτή την έκθεση ή τις εκθέσεις του κυρίου Γκέρες είναι επειδή είναι πραγματικά αδέκαστος ε, μας ρωτά και θέτει ερωτήσεις στους διαθρόμους, στο εστιατόριο, στα κηλικία αν έχει γίνει, αν έχουμε εξοικειωθεί με ε, έχουμε διαβάσει αυτές τις εκθέσεις ε, και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή, αυτό το έναυσμα. Πάντα είναι ενδιαφέρον ανάγνωσμα γιατί δεν, είναι, δεν αγνοούμε σε αυτή την Επιτροπή εκείνοι που είμαστε σε αρκετά χρόνια σε αυτό το έργο για το, το εύρος των γνώσεων και τις ικανότητες ε, του κυρίου Γκέρενς όταν στρέφεται σε αυτά τα θέματα που μελετά. Ήμουν μέλος και είμαι μέλος Επιτροπής, ιδιαίτερα και σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία και στην προηγούμενη όμως. Και συμμερίζομαι την ιδέα που εκφράστηκε ότι υπάρχει εδώ μια, ε, μια συνήθις πτυχή στις σχέσεις μα όταν έχουμε σχέσει για τι οποίε κάνουμε λόγο με χώρε που πρέπει να έχουν μαζί μας ένα διάλογο διαρθρωμένο, δομημένο, διαρκή, μόνιμο και αποτελεσματικό. Συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπε ο Νόρμπερτ πιο πριν ως προς το ότι αν γίνεται κάτι σε σχέση με τα πρακτικά τα οποία έχουν γίνει, αν τα μελετήσει κανείς και τις παρεμβάσεις στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές και σε σχέση με τις παρεμβάσεις στην ΑΚΕ υπάρχει μια μη ισόρροπη σχέση για το ενδιαφέρον που εκφράζουν τα, τα μέλη ΑΚΕ και το ενδιαφέρον που εκφράζεται σχετικά από τους ευρωβουλευτές. Έτσι εγώ θα θεωρούσα σκόπιμο λοιπόν, ώστε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση να είχαμε κάποιο είδους ανακοίνωση επίσημη ή ανεπίσημη προς τα μέλη, προς ε, τους, τα μέλη της ΑΚΕ που ανήκουν ως ευρωβουλευτές σε αυτήν, ώστε να αναφέρονται τα θέματα αυτά που θα εξεταστούν στο Στρασβούργο για παράδειγμα και οι παρεμβάσεις στο Στρασβούργο. Επιπλέον είναι καλή στιγμή να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε για ένα πλαίσιο σχέσεων με τις χώρες ΑΚΕ σε σχέση με ε, την ανάλυση που θα πρέπει να γίνει για το τι δεν λειτουργεί καλά και τι είναι εκείνο που πρέπει να αλλάξουμε για να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία, μια νέα κίνηση, μια νέα φάση οικονομικών σχέσεων για την ανάπτυξη. Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το έργο στο Ευρωκοινοβούλιο, την υποστήριξη δηλαδή σε σχέση με κάποιες χώρες της ΑΚΕ, ώστε να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στη διεθνή ε, σκακέρα, να διαδραματίσουν ένα ενεργό ρόλο, όπως για παράδειγμα για τον, ε, την ομάδα των, ε, την Λέσχη των 7 ή για του χρόνου το 2015, στους στόχους αυτούς ε, για το έτος ανάπτυξης το 2015 να συνδυαστούν οι προσπάθειες. Υπάρχει ένα σημαντικό μέρος αυτών των χωρών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην προσπάθεια νότου-νότου για την ανάπτυξη και σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία για την συνεργασία και την ανάπτυξη. Θέλω τέλος να επισημάνω ότι συμμετείχα σε πολλές συζητήσεις όπου εκφράστηκαν αμφιβολίες πολλές φορές για τις συμφωνίες εταιρικής σχέση αν πηγαίνουν καλά, μήπως ε, αναφέρονται σε μια ασυμμετρική σχέση ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε σε σχέση με τον ορίζοντα 2020 να αναθεωρήσουμε αυτές τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, και να δούμε αν θα το κάνουμε αυτό χώρα με χώρα ξεχωριστά ή στο διεθνές ε, πλαίσιο σφαιρικά ή αν πρέπει να συνεργαστούμε κάνοντας κάποια βήματα σε σχέση με κάποιες χώρες ώστε να ασκηθεί πίεση για παράδειγμα για οποιουσδήποτε λόγους που για τις πολιτικές τους αποφάσεις δεν πορεύονται προς αυτό το στόχο και δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον να μπορέσουν σε σχέση με την, ε, το πλαίσιο εταιρικής σχέσης να είναι αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς ζητήσατε να παρέμβετε για, ε, για την JPA, την Κοινή Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Θα θέλετε να παρέμβετε. I, Σημείωσα σε κάποιες συναντήσεις όπως της UNCTAD για την ε, ανάπτυξη ότι υπάρχει μεγάλη βούληση σε σχέση με τις χώρες ΑΚΕ αλλά ιδιαίτερα των αφρικανικών χωρών να συζητηθούν εναλλακτικέ δυνατότητες σε σχέση με αυτή την προσπάθεια. Και μάλιστα με, ήταν και επώδυνο αυτό διότι η διαδικασία επικύρωσης για παράδειγμα και όλες οι ε, δυνατότητες που δεν προχώρησαν λόγω διάφορων προβλημάτων πρόσβασης στην αγορά, ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην αγορά κτλ. Αυτό όμως που θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να εξετάσουμε είναι πώς οι αφρικανικές χώρες θα υποφελούνται, θα υποφελούνται από την υποστήριξή μας στις περιφερειακές ε, ενώσεις, ε, οργανώσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό, να αναπτύξουν δυναμικό αυτές οι επιχειρήσεις σε αυτό το περιφερειακό επίπεδο. Η ανατολικό-αφρικανική κοινότητα χωρών έναντι της δυτικο-αφρικανικής κοινότητας χωρών θα μπορέσουν να προαγάγουν λοιπόν το περιφερειακό εμπόριο από πλευράς τους Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την πτυχή και αυτή τη δυνατότητα και με το, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να τονωθούν αυτές οι προσπάθειες. Αυτό όμως έχει σχέση με το επόμενο θέμα, τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ ο κύριος Γκέρενς, αλλά όχι, ζητώ τον λόγο, ζητώ συγγνώμη Σαρλ, πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γκαμπέν, Χαμάν, εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε τον λόγο. Εντάξει όμως, πείτε μας το όνομά σας αν έχετε διαφορετικό όνομα, ποιος είστε. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Σαμάν θα μιλήσει για το επόμενο θέμα για τον ιδιωτικό τομέα. Σημερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν πολύ στις ανησυχίες και τις διαπιστώσεις της έκθεσης αυτής ότι δηλαδή υπάρχει κάποια θα έλεγα αδυναμία στην ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στους χώρους αυτούς. Για μας ε, αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο συνάντησης, πρόκειται για κάτι το οποίο θα επιτρέψει μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, περισσότερο σε περιφερειακό επίπεδο, παρά σε επίπεδο ολομέλειας όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο επίσημα και τυπικά. Δεν έχουμε αντιρρήσεις λοιπόν κάποια σε επίπεδο συντακτικά θέματα περισσότερο, σε επίπεδο συντακτικό. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να στέλνει γραπτές απαντήσεις στις προφορικές ερωτήσεις οι οποίες κατατίθενται ε, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του JPC. Να πω εδώ ότι οι προφορικές ερωτήσεις απαντώνται προφορικά. Αλλά βέβαια φυσικά και δεχθήκαμε εδώ και αρκετά χρόνια να δίδουμε και γραπτές απαντήσεις στους βουλευτές εκ των προτέρων, κάτι το οποίο επιτρέπει κατά τη διάρκεια της συζήτησης να μην παραμένει κανείς παρά στα θέματα τα οποία είναι ε, σε εκκρεμότητα. Θα ήθελα όμως να πω ότι αυτή η δυνατότητα την οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το Συμβούλιο παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες γιατί στα πλαίσια αυτής της προαιρετικής μας πρωτοβουλίας είδαμε ότι χαρακτηρίζεται μονομερός στο άρθρο 21 των κανονισμού και μιας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δεσμεύεται από τους κανόνες αυτούς, θα θέλαμε να ζητείτε η άποψή μας στα πλαίσια της Διοργανικής Συμφωνίας Κοινοβουλίου Επιτροπής. Αλλά για να τελειώσω μια θετική παρατήρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να δίδει γραπτές απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στον φίλο Γκουερέρο ότι δεν κατηγορώ αυτούς που δεν διάβασαν την έκθεσή μου. Υπάρχουν εκθέσεις πολύ που ενδιαφέρουσες. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζει κάποια ενδιαφέρον. Μπορώ να τους δώσω και μία περίληψη σε αυτούς οι οποίοι δεν την έχουν διαβάσει. Ο κύριος Πόγκας σωστά Διαρωτάτε το τι θα γίνει μετά το 20. Θα πρέπει ήδη να το λάβουμε υπόψη μας. Η συνέχεια μιας πολιτικής, η, η ρήξη μιας πολιτικής πρέπει να αποφασίζεται νωρίτερα μέσα στο χρόνο. Είναι θετικά πάντως τα αποτελέσματα στα οποία έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα και εδώ θα σας στηρίξω πλήρως. Από κοινού με τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη θυμίζω ότι δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις μας ενώ έχουν κάθε δυνατότητα να το κάνουν αν το επιθυμούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει μετά το 2020 από κοινού. Δεύτερον, πολλές ερωτήσεις ασχολούνται με το πώς μπορούμε να εκδημοκρατήσουμε περισσότερο τη λειτουργία των ΑΚΕ. Αναφέρθηκε η διαδικασία και χωρισμένης ψηφοφορίας. Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή είναι αρκετά περίεργη θα έλεγα και ανταποκρίνεται στην δημιουργία της σχέσης ε, με τις χώρες ΑΚΕ. Δεν μπορούσαμε μονομερός να πάρουμε μια κάποια απόφαση και γι' αυτό προτείνουμε τη συγκεκριμένη λύση. Στα πλαίσια τώρα του εκδημοκρατισμού της διαδικασίας να αναφερθούμε στο θέμα του δημοσιονομικού ελέγχου. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ε, κάποιες αρμοδιότητες καθαρά δημοσιονομικές οι οποίες κανονικά ανήκουν σε μια κοινοβουλευτική συνέλευση. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να δράσουμε καλύτερα από ό,τι το κάνουμε μέχρι τώρα. Είχα θέσει το ερώτημα στον τέος επίτροπο τον κύριο Πίμπαλξ για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ο ίδιος συμφωνούσε να πάει στα κοινοβούλια των κρατών μελών και να παρουσιάσει το θέμα. Το μόνο κοινοβούλιο το οποίο είχε ζητήσει την δυνατότητα αυτή ήταν το κοινοβούλιο της Μπουρκίνα Φάσο. Κανένα κοινοβούλιο από τα κράτη-μέλη της Ένωσης δεν είχε ζητήσει την παρουσία του. Οπότε και εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Σε συνεργασία με τα κοινοβούλια των χωρών μας μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα ε, και θα το συζητήσουμε το θέμα στην επόμενη συνάντηση. Αν υπάρχουν τόσοι λίγοι υπουργοί παρόντες στις συνεδριάσεις ε, με τις χώρες ΑΚΕ, αυτό συμβαίνει γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έρχονται ποτέ. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν υπουργού σε θέματα ανάπτυξης και ακόμα και αν έχουν δεν συμμετέχουν συχνά ε, στις υπουργικές ε, ε, συναντήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο επιφυλακτικοί αντικαθιστώντας αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτές τις συναντήσεις από πραγματικά πολιτικούς υπευθύνους. Όταν έγινε η τελευταία συνάντηση στον Κόγκο, η Υπουργή Ανάπτυξης, ο Υπουργός Ανάπτυξης του Βελγίου τότε δεν είχε την δυνατότητα να αντικαταστήσει ε, την ευρωπαϊκή πλευρά. Υπήρχε ένα θέμα λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπηθούν τα κράτη-μέλη σε πολιτικό επίπεδο το όργανο το κοινοβουλευτικό αυτό δεν είχε την δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις που μένει να γίνουν λοιπόν και ο συντονισμός των πολιτικών θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο από όσο μέχρι τώρα. Τέλος, νομίζω ότι η κυρία Χάουταλα το έθεσε αυτό. Αναφέρομαι στις συμφωνίες ε, οικονομικής ε, συνεργασίας που αποφασίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο περιφερειακών διασκέψεων. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να δούμε τι θα γίνει και με τις επιπτώσεις του TTIP για την Αφρική, για τις χώρες ΑΚΕ. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε καταθέσει τις τροπολογίες σας. Ε, παρακαλώ να το κάνετε. Ευχαριστώ Σαρλ. Το θέμα της ψηφοφορίας πραγματικά δείχνει ακριβώς τι είδους προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. πώς μπορούμε να εμφυσίσουμε περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα, όπως είπε και ο κύριος Μασκούρ στη συνέλευση με τη ΣΑΚΕ. Λοιπόν, φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα, περνάμε τώρα στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Για τον ιδιωτικό τομέα αποφασίσαμε να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας, ιδίας πρωτοβουλίας, DIVA. Δεν έχουμε κείμενο. Θα ακούσουμε τον εισηγητή, θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημοσίευσε και μία έκθεση για ένα ισχυρότερο ρόλο στον ιδιωτικό τομέα πριν από τις τελευταίες εκλογές και γι' αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της χρηματοδότησης ε, για την ανάπτυξη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντίβα και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση και έχω ήδη τον κατάλογο των σκιωδών και δεν ξέρω ποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους. Έχω πει πολλές φορές σε αυτή την Επιτροπή πόσο σημαντικό είναι τα κονδύλια μας να δημιουργούν πλούτο και ανάπτυξη. Η ε, ανακούφιση της φτώχειας μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με δημιουργία πλούτου. Πόσο σημαντικό είναι για τις αναπτυξιακές πολιτικές να στηρίζονται στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα πόση σημασία έχει ο κόσμος στις ομένες χώρες ε, να έχει πράγματα στην ιδιοκτησία του, να μπορεί να ανοίγει μια επιχείρηση σε μέρες και όχι και χρόνια και να λειτουργεί στην επίσημη οικονομία. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ο κινητήρας της ανάπτυξης σε όλες τις οικονομίες της αγοράς. Δημιουργεί το 90% των θέσεων της εργασίας και του εισοδήματος και βεβαίω κινητοποιούνται έτσι οι εσωτερικοί πόροι για να αναπτυχθούν οι χώρε. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για την ανακοίνωση αυτή τη Κομισιόν για τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Υπό την ηγεσία του πρώην επιτρόπου του κυρίου Πίμπαλξ, η Κομισιόν δικαίω τονίζει τρεις τομείς στου οποίου μπορούμε να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ειδικά η ενδυνάμωση της ζωής των γυναικών ε, σε όποιο πολιτισμό και αν ζουν. Γεγονός είναι πως μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να ε, αντιμετωπίζονται ως ίσες. Και μετά περνάμε στους άνεργους και στους φτωχότερους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε της, ε, το επιχειρησιακό περιβάλλον, την πρόσβαση στην χρηματοδότηση για να προωθήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες συχνά αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα ρυθμιστικά εμπόδια συχνά λειτουργούν ε, στην ε, ανεπίσημη οικονομία και δεν έχουν νομική προστασία. Οι κανονισμοί που υπάρχουν διώχνουν τις μικρές επιχειρήσεις και τις οθούν στην ανεπίσημη οικονομία. Εκατομμύρια τέτοιες ε, στους δρόμους όπως κανείς πηγαίνει από το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα. Υπάρχει κόσμος που μαστορεύει πράγματα, κατασκευάζει πράγματα αλλά δεν είναι στην επίσημη οικονομία, δεν μετράνε στο ΑΕΠ. Δεν μπορούν να πουλήσουν και να, να και να αγοραστούν οι επιχειρήσει. Δεν έχουν καμία αξία παρά μόνο γιατί δεν έχουν κάποια αξία. Ε, δεν υπάρχει ε, δεν υπάρχουν λογιστικά βιβλία, έσοδα, έξοδα, δεν είναι καταγεγραμμένες ως εταιρείε, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις. Στι αναπτυσσόμενες χώρε. Και είναι όλες στον ανεπίσημο τομέα. Αν περάσουν στην επίσημη οικονομία, το ΑΕΠ των χωρών αυτών θα εκτοξευτεί. Επίσης, περιβάλλον φιλικό για την ιδιωτική πρωτοβουλία και το να μπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επίσημη οικονομία πρέπει να είναι προτεραιότητα μαζί με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δεύτερον, μπορούμε να συνεργαστούμε με τον διεθνή ιδιωτικό τομέα. για να έχουμε ακριβώς βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σοκαριστικό ότι 51 από τις 100 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο είναι επιχειρήσεις. 51 από τις 100 είναι επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες 500 πολυεθνικές είναι γύρω στο 70% του παγκοσμίου εμπορίου. Τεράστιο δυναμικό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αν συνεργαστούμε μαζί τους. Και τεράστια ευθύνη. Μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τους για να μειώσουμε τη φτώχεια. Αλλά σήμερα δεν είμαστε σε επαφή μαζί τους στην Επιτροπή αυτή. Και παρόλες τις καλές μας προθέσει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν ακούσουμε και δεν μιλήσουμε και δεν συνεργαστούμε με το τι έχει να πει το 51% των μεγαλύτερων παγκοσμίων οικονομιών. Ε, δηλαδή τι λογική είναι αυτή. Όλο και περισσότερες από αυτές τις εταιρείες συνειδητοποιούν πως συνεισφέρουν ε, με το να λειτουργούν ε, με τρόπο ώστε να βοηθούν την ανταγωνιστικότητα, να βοηθούν το περιβάλλον και τις κοινωνικές προδιαγραφές. Μπορούμε μαζί τους λοιπόν να αναπτύξουμε επιχειρηματικά μοντέλα που θα ενσωματώνουν τους φτωχούς είτε ως υπαλλήλους διανομής και τα λοιπά, γιατί οι εταιρείε αυτές χρειάζονται αυτές τις δεξιότητες. Είναι προς το συμφέρον αυτών των εταιριών να βελτιώσουν τις δεξιότητες των φτωχών. Γιατί το τα, τους χρειάζονται. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουν στην αλυσίδα της προσθέμενης αξίας, είναι λοιπόν αμοιβαία αποφελές αυτό. Και για όσους θέλουμε να επιτευθούν οι στόχοι της χιλιετίας και να καταπολεμηθεί η φτώχεια και για τις εταιρείε που θέλουν πιο ειδικευμένους εργαζόμενους ε, για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Τρίτον, υπάρχει ο τομέας της γεωργίας, ε, της υγείας, η έρευνα και ο πράσινος τομέας συνολικά. Όταν μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ε, πείρα και τα συστήματα και τα συστήματα διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα γνωρίζουν πώς να το κάνουν, έχουν αυτό το δυναμικό. Γιατί δεν τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε να μπορέσει αυτό να αποβεί προς όφελος όλων των φτωχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μας, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας. Υπάρχει αυτή η πραγματογνωμοσύνη, οι γνώσεις σε εταιρική σχέση με τους ε, κοινούς πόρους. Ο ιδιωτικός τομέας συνεισφέρει σημαντικά ήδη ώστε να <clears throat> μπορεί να παρέχεται ασφαλές ε, νερό για πόση παγκόσμια, για την ανάπτυξη αγορών, για την ε, η ανάπτυξη ιδιωτικών δημόσιων σχέσεων. 34 δις δολάρια τα τελευταία 10 χρόνια δεν θα μπορούσαν να εξευρεθούν αυτά τα 34 δις ε, για πόσιμο νερό για να παρέχεται στους φτωχούς. Ο ιδιωτικός τομέας μπόρεσε να τα βρει αυτά τα ποσά. 34 δολάρια ώστε να μπορούν να έχουν αυτά τα ε, το αγαθό αυτό, το πόσιμο νερό αυτοί οι πληθυσμοί, να μπορούν να πίνουν καθαρό νερό την πατρίδα τους. Έχουμε λοιπόν αυτή την προοπτική. Οι ιδιωτικές εταιρείες, οι περισσότερες, δεσμεύονται νομικά να παρέχουν διαφανές πλαίσιο των εργασιών τους και να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε μεγάλο βαθμό οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο διαφάνειας. Έτσι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους ώστε να ενθαρρυνθεί η χρηστή διακυβέρνηση και διαχείριση μέσα σε ένα πλαίσιο κράτους δικαίου, ρύθμιση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, καταπολέμηση διαφθοράς και να μπορέσει έτσι λοιπόν πραγματικά στον τομέα των περιφερειακών και των τοπικών να αναπτυχθεί αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία. Πολλά πρέπει και μπορούν να γίνουν. Χρειαζόμαστε τις ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, τους εμπλεκόμενους, τις κοινέ ε, κοινοτικές αρχές, ε, δημοτικές αρχές, δήμους, κοινότητες, τοπικά και περιφερειακά να συνεργαστούν όλοι προς όφελος των φτωχότερων στις χώρες και στις περιοχές αυτές, ώστε με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις ε, για να υπάρχει δικαιοσύνη και σωστή λειτουργία και διακυβέρνηση οι φτωχοί να έχουν μια δυνατότητα να έχουν λίγα περισσότερα χρήματα, να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση, να συμμετάσχουν, να δημιουργηθούν αξίες και πλούτος. Και αυτές είναι οι φιλοδοξίες μας και γι' αυτό την επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών χρειάζομαι την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γκαμπέν Χαμάν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ σας ζητώ να μας δώσετε πληροφορίες και επικοινωνικά, επικοινωνιακά σχετικά με αυτά. Σε σχέση με το, τους στόχους σας, ε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πώς αξιολογείτε το έργο αυτό από πλευρά σας. Εσείς παρακαλώ, έχετε λοιπόν τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ε, ο συνάδελφος Βιναμάν δίπλα μου κάθεται. Ε, σας, καλώς, σας Εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους σας. Έχετε πολύ απόλυτο δίκιο ότι πολύ λίγα μπορούν να προσθεθούν πρόεδρε σε αυτά που είπε ο αξιότιμος Ευρωβουλευτής Νίρτς Ντέβα. Αυτές είναι οι αρχές, οι κύριες δυνάμεις πίσω από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτό το στόχο. Κάποιες παρατηρήσεις να κάνω μόνο για να συμπληρώσω αυτή την παρουσίαση και μετά να πω προς τα που κινούμαστε από αυτό το σημείο. Οι αρχές και τα κριτήρια αυτής της εμπλοκής με τον ιδιωτικό τομέα είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό και πολύ καλά εξηγείται, επεξηγείται στην ανακοίνωσή μας. Όχι μόνο έχουμε αυτό το οποίο απαρίθμησε ο κύριος Ευρωβουλευτής Νίρς Ντέβα για τις συνέργειες τους συνδέσμους και τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, την καινοτομία που μόνο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να, ασφαλί, να εξασφαλίσει και για την απασχόληση και δράση, αλλά επίσης αυτά που είναι η διαδραστική, το διαδραστικό πλαίσιο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πώς και οι δημόσια κονδύλια μπορούν με, τους, ε, τα ιδιωτικά κεφάλαια να συνεργαστούν. Πολύ μεγάλη σπουδαιότητα σε αυτό το σημείο. Θα έχουμε μόχλευση και μοχλευτικό αποτέλεσμα από αυτές τις δράσεις. Σίγουρα ναι. Και θέλουμε οπωσδήποτε να αποφασίσουμε με ποιους τρόπους, με ποιες αρχές θα γίνεται αυτή η αμφίδρομη δράση. Αυτές οι αρχές μπορούν και με κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εκπορεύονται. Οδηγίες για τη διαφάνεια και πρωτοβουλίες που είχαν αναλυφθεί κατά το παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από αυτά είναι το φλέκτα, η επιβολή του νόμου για την διακυβέρνηση και το εμπόριο. Η αρχή αυτή αποτελεί κάτι το πολύ σημαντικό για την διαδραστική αμφίδρομη δράση ιδιωτικού ε, τομέα και ε, δημοσίων πρωτοβουλειών. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν το σωστό ρόλο που θα αναλαμβάνουν. Ας το αναφέρουμε αυτό ρητά και κατηγορηματικά και με τις, ε, τους συνεταιρισμούς εταιρική σχέση να το πούμε θέλουμε να προαγάγουμε με την παραγωγή στην γεωργία ώστε να μπορέσει να αναβαθμιστεί το έργο των γεωργών που δεν είναι μόνο παροχή τροφής αλλά δίνοντας και τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται τα παιδιά και να μπορούν μετά να παρακολουθούν ε, οι νέοι μαθήματα σε πανεπιστήμια να αναβαθμιστεί η δραστηριότητα όχι μόνο να παράγουν τρόφιμα για διατροφή αλλά να υπάρχει και η περαιτέρω ανάπτυξη να διασυνδέσουμε την καινοτομία στην έρευνα για τη γεωργία ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε και να δημιουργήσουμε μεγάλο πλούτο, πολυσχηδός, πράγμα το οποίο θα είναι εποφελές. Δεν θέλω να προσθέσω πολλά πράγματα. Έχουμε 12 δράσεις που απαριθμούνται στην ανακοίνωση στο, στον τομέα πολιτικής ρυθμιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης πολύ συχνά κάνουμε λόγο για τη χρηματοδότηση Μεγάλο πλαίσιο χρηματοδότησης είναι διαθέσιμο για τους ιδιωτικούς επενδυτές. Πολύ συχνά δεν είναι όμως το σωστότερο πλαίσιο. Έχουμε πολλούς ε, κανόνες και κανονισμούς με πολύ ψηλά επιτόκια και ε, πολύ στενές ε, προθεσμίες για την απόσβεση. Χρειάζονται όμως χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερο χρόνο απόσβεσης. Αυτή η αποτυχία λοιπόν στην αγορά πρέπει να αλλάξει. Έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Η Τη της υπαίθρου τεράστια σημασίας. 500 εκατομμύρια νέες συνδέσεις ηλεκτρικές ε, για σπίτια και νοικοκυριά προσιτή ενέργεια και σε προσιτές τιμές για όλους. Αυτό είναι ο συσχετισμός σε σχέση με την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση στα, ενεργειακά προϊόντα και πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούμε και να επενδύσουμε και μέσα σε ένα πλαίσιο μ, κινδύνων να αυξήσουμε την αηφορία. Έχουμε λοιπόν τις προτάσεις αυτές ε, για προσέγγιση ΜΚΟ, όμως η αηφορία ενός ιδιωτικού επενδυτή, μιας ιδιωτικής ε, ε, εταιρείας που εξετάζει τη σύνδεση πολλών ε, πολιτών με το ηλεκτρικό ρεύμα με την ηλεκτρική ενέργεια είναι θετικό γιατί θα δοθεί ευκαιρία να επιτευχθεί αυτό υπό τους ε, πιο σωστούς όρους. Ανοίγουμε εταιρική σχέση μεταξύ ΜΚΟ και μικρών επιχειρήσεων, πολύ μικρών επιχειρήσεων που θα επενδύουν στην Ήπεθρο. Αν περιμένουμε να υπάρξουν τα μεγάλα έργα, μεγάλες, ε, μεγάλη αγωγή για να λειτουργήσουν όλα αυτά, σε 50 χρόνια θα φτάσουμε στους πολίτες που έχουν ανάγκη να συνδεθούν. Πρέπει άμεσα να υπάρχει σύνδεση με προσπελάσιμο ε, εύκολο τρόπο πρόσβασης. Γι' αυτό πρέπει να επιτευχθούν οι επενδύσεις. Πολλοί επενδυτές και επιχειρηματίες δεν είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε ένα επικίνδυνο για τα κεφάλαιά τους περιβάλλον στην υποσαχάρη Αφρική. Και αυτό είναι μια αποτυχία πάλι. Ας το πούμε κάθετα και ξεκάθαρα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την αποτυχία και αυτό το πρόβλημα να το άρουμε για να είμαστε επιτυχείς. Θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε. Το mainstreaming, ένταξη όλων αυτών των αρχών δηλαδή και των κριτηρίων στις πολιτικές μας. Ένταξη όλων αυτών των δράσεων που σας προανέφερα στους τομείς εκείνους που τόσο εύλογα και με τόσο ε, θα έλεγα επιτυχή ρητορία εν τη ρήμη του λόγου του εξέθεσε ο κύριος Νίλς Ντέβα για την ανάπτυξη της εμπορικής ειδικού χαρακτήρα γεωργίας έχουμε πολύ καλές εταιρείες που μπορούν να αναπτυχθούν και πρέπει να αναπτυχθούν. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση του πληθυσμού πρέπει να επιτευχθεί. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό πάντα. Αυτές τις αρχές ε, για αυτή την ανάπτυξη θέλουμε να τις αναπτύξουμε με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να πετύχουμε μόχλευση. Μόχλευση στις παραγωγικές επενδύσεις για την ανάπτυξη. Συνεισφέροντας ώστε αυτές ε, οι δράσεις από άτυπο πλαίσιο να μετατεθούν, να μεταφερθούν σε ένα επίσημο, επισημο, επισημοποιημένο πλαίσιο για την οικονομία. Αυτό θα κινητοποιήσει το δυναμικό ώστε να επιτευχθούν επενδύσεις ε, όπως πρέπει. Δεν γνωρίζω πρόεδρε, απάντησα συνολικά σφαιρικά στο ερώτημά σας, στα ερωτήματά σας. Το μέλημά μας είναι στον προγραμματισμό δια ΑΚΕ μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και των διαφορετικών δράσεων γεωγραφικά, τομεακά και κλαδικά να εξεύρουμε εκείνου τους τομεί αναφέρθηκαν δύο η ενέργεια και η γεωργία και οι αγροεπιχειρήσεις όπου η ανάπτυξη μέσω του ιδιωτικού τομέα και όταν λέμε ιδιωτικό τομέα λέμε μικρές, αναφερόμαστε σε μικρές και μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν κάνουμε λόγο για πολυεθνικές και ελπίζουμε ότι αυτές οι επενδύσεις θα επιτευχθούν μέσω των προσπαθειών μας και θα υπάρξει πολλαπλασιασμός αυτών των ε, προσπαθειών. Δεν υπάρχει αρκετό κακάο για παράδειγμα για την σοκολατοβιομηχανία της Ευρώπης. Ο μόνος εφικτός και αηφόρος τρόπος είναι να αυξηθούν τα κονδύλια ώστε να καλλιεργούν κακαόδεντρα στην Αφρική η Διαφορετικά δεν θα υπάρξει επαρκής παραγωγή σοκολάτα στην Ευρώπη. Είμαι πρόθυμος να ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Έχουμε όμως σαφή κινητήρα, σαφή παράμετρο για την κινητήριο δύναμη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις επενδύσεις που χρειάζονται. Ζητούμε στη, να εμπλακεί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και έτσι θεματολογικά θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις διαφορετικές μας δράσεις πολύ συχνά εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα στην ηλεκτροδότηση, στη δράση ηλεκτροδότησης της υπαίθρου που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οι εξή έχουν ζητήσει το λόγο. Στιερ, Νόιζα, Άουταλα, Γκέρεντς και Σίλβα Περέιρα και Σάντσες. Θέλει κάποιος άλλος και Γκουερέρο. Και εγώ άλλωστε. Τρία λεπτά ο καθένας. Νταβόρ. Θα είμαι σύντομος πρόεδρε. Πρώτον, να ευχαριστήσω τον ΕΡΖ για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις και για την ευκρίνεια του μηνύματός του. Να ευχαριστήσω και τον πρέσβη κύριο Ριντόλφη, ο οποίος είναι πράγματι ένα παράδειγμα αντίθετο με την εικόνα που έχουμε για τους ε, γραφειοκράτες, ένας άνθρωπος που έχει πάθος και το πάθος έρχεται από την εμπειρία του στις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, όλα συνδέονται με τις αγορές. Μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να αφήσουμε τα πράγματα να εξελίσσονται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ή μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η αγορά αποτυγχάνει και υπάρχει ανάγκη για καλύτερη και ευρύτερη διακυβέρνηση και είναι απαραίτητο λοιπόν να ξεκινήσει ο διάλογος αυτός με τον ιδιωτικό τομέα. Μπορούμε να επανέλθουμε στα θέματα αυτά με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Νόιζα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Ντέβα. Νομίζω κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να τα πει πιο καλά για τον ιδιωτικό τομέα και τις δυνατότητες της αναπτυξιακής ε, πολιτικής. Νομίζω πρέπει να δούμε αυτό το θέμα πιο ρεαλιστικά και λιγότερο ιδεολογικά. Παρόλα αυτά θέλω να κάνω μια παρατήρηση που είναι σημαντική για εμάς τους σοσιαλδημοκράτες. Γιατί πρέπει νομίζω να οδηγηθούμε σε καλή επιχειρηματική πολιτική, κάτι το οποίο σημαίνει βεβαίω και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία λογική ε, ανάπτυξη Επίσης, οι γυναίκες. Πρέπει να σκεφτούμε και τους νέους. Η Αφρική είναι πάρα πολύ νέα ήπειρος με αρκετά μεγάλο δυναμικό και όπου ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα σε πολλές χώρες όπου η νέα γενιά εργάζεται δημιουργικά και βεβαίως πρέπει να τη στηρίξουμε. Τρίτον, η Κομισιόν πραγματικά έκανε καλή δουλειά και ακριβώς αυτό είναι το θέμα που, είχα, που λέω πάντα στην αναπτυξιακή πολιτική. Χωρίς μια λογική ε, πολιτική ενέργειας δεν γίνεται τίποτα. Αν κάποιος είναι ε, χειρόναξε, 6 ώρα το απόγευμα τελειώνει η δουλειά του γιατί δεν έχει φως. Ένα παράδειγμα λοιπόν που δείχνει πως χρειαζόμαστε αηφόρο ε, ενέργεια σε περιφερειακό επίπεδο για να, αναπτυχθεί, για να αναπτυχθούν οι χώρες αυτές. Ε, ευχαριστώ. Χάουταλα και μετά Σαλ Γκέρενς. Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε πρέπει να συνεισφέρει ο ιδιωτικός τομέας και θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω κάποιες ιδέες. Αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν βεβαίω είναι πάρα πολύ θετικό και θα ήθελα και εγώ να το επαναλάβω το θέμα δεν αφορά τις πολυεθνικές αλλά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το να δημιουργηθούν νομίζω νέε θέσει εργασία γιατί δεν υπάρχουν δουλειέ, ε, είναι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τη βάση τη λεγόμενη της πυραμίδα. Πώ μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε τους φτωχότερους να μπορούν να συντηρηθούν. Ακόμα και στις λεγόμενες, ε, στα λεγόμενα, λεγόμενες παραγκουπόλεις. και βλέπουμε πως οι ακτιβιστές, οι πανεπιστημιακοί έχουν βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να βγάλουν το βιός τους. Έχουμε πολλά νομίζω να κάνουμε στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης γιατί όπως είπε ο κύριος Νόιζερ υπάρχουν νέοι που πρέπει να πάνε ε, δημοτικό και γυμνάσιο και να μάθουν και κάποια τέχνη. Και βεβαίω κάποιες μεγαλύτερες εταιρείες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν εδώ πέρα στην επαγγελματική κατάρτιση γιατί συχνά ακριβώς ε, δεν υπάρχουν ε, οι δυνατότητες για να δουλέψει κάποιος ε, στην βιομηχανία. Η τεχνολογία είναι σημαντικό, αναφέρθηκε ήδη πρόσβαση στην ενέργεια. Θυμόμαστε πως ο Μούν εξήγησε πως ε, δεν μπορούσε ούτε καν να διαβάσει όταν έδιε ο ήλιος γιατί δεν υπήρχε καν φως. Ε, πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε το 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που δεν έχουν ρεύμα να αποκτήσουν. θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως οι περισσότεροι φτωχοί άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η βασίλισσα της Ολλανδίας ε, έχει αφιερωθεί στο να βοηθάει τους φτωχούς να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Οπότε πολλά μπορούμε να, για το, να πούμε για το τι μπορεί να γίνει για τους στοχούς και βεβαίως η άλλη διάσταση είναι οι υποχρεώσεις των διεθνών εταιριών. Γνωρίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά παρουσιάζεται ως ε, εκείνη η οποία προστατεύει τους μεγάλους επενδυτές. Τι γίνεται όμως με τις υποχρεώσεις και ερχόμαστε εδώ πέρα στους κανόνες για την ε, κοινωνική ευθύνη. Και βλέπω πως ε, πηγαίνουμε προς δεσμευτικούς κανόνες. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Πρέπει να δημιουργηθούν ίσοι κανόνες ανταγωνισμού. Η Κομισιόν ανέφερε κάποιες σωστές πρωτοβουλίες, Φλεκτ, πράγματι και άλλες και το EITI για τις εξορρυκτικές ε, βιομηχανίες που πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία για να μπορούν και οι χώρες αυτές να ε, παίρνουν κάποια από τα κέρδη των εξορρυκτικών εταιριών και βεβαίως θα μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται και με τους ανανεώσιμους πόρους όπως τα δάση, το κυνήγι κτλ. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. και νομίζω πρέπει να συνεισφέρουμε στη δουλειά του ε. κύριου Ντέβα. Ευχαριστώ. Σαλ Γκέρνς και Πέντρο Σίλβα Ευχαριστώ. Οι εκθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες αυτές, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μας δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν ξεφύγει. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χωρών στην Αφρική που έχουν απογειωθεί με οικονομικούς ρυθμούς ανάπτυξης 10% σχεδόν. Κάποιοι φτάνουν στην Γκάνα, ας πούμε, 14%. Το θέμα είναι αν η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί μέσα καταπολέμησης της φτώχειας. Πράγματι ε, παράγεται πλούτος, αλλά χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της φτώχειας. Δυστυχώς όχι ένα καινούριο πρόβλημα. Τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να πιέσουμε. Τι μία, έχουμε την έννοια της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την καινούργια πολιτική ανάπτυξης. Η έννοια αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, γιατί στα πλαίσια αυτής της πολιτικής έχει σημασία να ε, χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας αποκλειστικά για αυτούς τους στόχους, γιατί αλλιώς τότε θα βγούμε εκτός των ε, προοπτικών ανάπτυξης. Αν θέλει να αναπτύξει κανείς τη βιοτεχνία σε μια χώρα, είτε μπορεί να το κάνει ε, στα πλαίσια του στόχου καταπολέμηση της φτώχειας, οπότε θα πρέπει να καταρτήσει τους νέους που δεν έχουν καμία γνώση και δυνατότητα για να τους βγάλει από τη φτώχεια και να τους δώσει προοπτικές. Αν στα πλαίσια της αναφοράς επιμείνει στην απαραίτητη λοιπόν προσπάθεια κατάργησης της φτώχειας, τότε αυτός ο οποίος θέλει να πετύχει είναι ακριβώς αυτό το οποίο προτείνουμε. Ή αλλιώς δεν διευκρινίζει κανείς την καταπολέμηση της φτώχειας στους όρους αναφοράς και αναπτύσσει τον τομέα προωθώντας αυτούς οι οποίοι είναι ικανότεροι. Δύο ακραία παραδείγματα. Στο πρώτο παράδειγμα η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη είναι αναπόσταστο τμήμα του συστήματος. Στο δεύτερο παράδειγμα παίζει δευτερεύοντα ρόλο Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορέσουμε να προσμετρήσουμε εμείς τις επιπτώσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ήδη είναι σε θέση να μας δώσει ένα μας σύντομο το οποίο να ε, επηρεάζει, να δείχνει πόσο επηρεάζουν τα μέτρα μας στην πολιτική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ε, στις χώρες οι οποίες παίρνουν τα χρήματα τα κοινοτικά. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τη λεγόμενη αρχή της διαφοροποίησης. Εμείς στηρίζουμε τις χώρες οι οποίες έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και δεν μπορούν μόνες τους να διασωθούν και αποχωρούμε από τις χώρες οι οποίες μπορούν να, ε, με δικά τους μέσα να καταπολεμήσουν την ε, φτώχεια. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό για να δείξουμε ότι οι αρχές έχουν ε, μέσα τους ένα βαθύτερο νόημα και το νόημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Όλες οι διασκέψεις που έχουμε μπροστά μας πρέπει να καλύπτουν τις ε, σημαντικές ε, μορφές εφαρμογής αυτών των βασικών αρχών εφόσον επιθυμούμε να πετύχουμε. Έχουμε το παράδειγμα το λατινοαμερικανικό το οποίο παράγει πλούτο και φτωχούς ταυτόχρονα ή θα ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε ακριβέστεροι. Εγώ δεν κατηγορώ εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή της συγκεκριμένη αρχής. Σας ευχαριστώ. Σίλβα σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο συνάδελφός μας Ντέβα Νίρτζ έθεσε τις σωστές βάσεις για τη συζήτησή μας για αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Και θα ήθελα να πω επίσης εγώ ότι καθώς ε, είχαμε το θέμα της προετοιμασίας της έκθεσης για μετά το 2015, χωρίς αμφιβολία αυτό το εγχείρημα για τη δράση του ιδιωτικού τομέα θα έχει ένα σημαντικό input. Σημαντικές προτάσεις θα απορρεύσουν για τη δουλειά που πρέπει να γίνει για την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μετά από το 2015. Αυτό που του οποίου πρόκειται, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, είναι κάτι παραπάνω από την παραδοσιακή ε, ευθύνη επιχειρήσεων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αφενός να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε ώστε η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα στις οικονομίες υπό ανάπτυξη χωρών είναι μία συνεισφορά αυτονόητη για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της διαδικασίας της, των διαδικασιών της ανάπτυξης. Αλλά όχι μόνο η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα είναι ο αναγκαίος όρος. Γι' αυτό οι αρχές, οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα συνεισφέρουν για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα είναι σημαντικά θέματα. Υπογραμμίστηκε και συμφωνώ απόλυτα για το ρόλο της διαφάνειας π.χ. Το ρόλο που έχει η διαφάνεια όμως η καταπολέμηση της παραοικονομίας δεν είναι μόνο ένας τρόπος να έχουμε την σωστότερη απεικόνηση της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας. Είναι επίσης ένας τρόπος να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Διότι όταν έχουμε μια οικονομία που είναι παράλληλη οικονομία σε σχέση με την επίσημη οικονομία που επιβάλλει φόρους Κανένα μέσο επιμερισμού πλούτου στην οικονομία και καταπολέμησης της φτώχειας δεν μπορεί να δώσει καρπούς. Γι' αυτό είναι ένας όρος για τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα η καταπολέμηση της παραοικονομίας. Επίσης, όσον αφορά την ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα με τους στρατηγικούς στόχους της ανάπτυξης που πρέπει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Είναι μια πολύ σημαντική πτυχή και αυτή που μας οδηγεί στα μέσα και τα εργαλεία για τις σχέσεις. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πείρα για την χρήση και την του τι συμβαίνει στις εταιρικές σχέσεις δημόσιες ε, και ιδιωτικές. Ενδιαφέρον θα ήταν να αναπτύξουμε την πρόταση των πολιτικών για την ανάπτυξη με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει παιδαγωγικός ρόλος ε, για την χρήση αυτών των ε, μέσων και εργαλείων στην εταιρική σχέση δημόσια και ιδιωτική. Και τέλος, για τους ίδιους τους όρους χρηματοδότησης. Χρηματοδότησης της ανάπτυξης μέσω ακριβώς των προσπαθειών για τον ιδιωτικό τομέα, της πρόσβασης ε, όσον αφορά κοινοτικά κονδύλια, άλλα κονδύλια που είναι διαθέσιμα επίσης και τους όρους ε, δανειοληπτικής δυνατότητας, διάθεσης πιστώσεων. Αυτό είναι σημαντικό, είναι σφάλμα να σκεφτούμε το μέλλον της πολιτικής για την ανάπτυξη χωρίς να δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα διαφυλάσσοντας τις αναγκαίες αρχές που πρέπει να διαφυλαθούν το ρόλο που πρέπει να διασφαλίσουμε στον ιδιωτικό τομέα. Θα ήταν σφάλμα να τα αγνοήσουμε αυτά. Ευχαριστώ. Λόλα Σάντσες και ο Ενρίκε Γκερέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς σε σχέση με τον αισιόδοξο, την αισιόδοξη αντιμετώπιση του ιδιωτικού τομέα έχουμε διαφοροποιημένη θέση. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας και ρήτρε ασφαλείας που θα δίνουν τη δυνατότητα ο ιδιωτικός τομέας, το ιδιωτικό κεφάλαιο να μην υπονομεύει την πρόοδο και τις δυνατότητες ανάπτυξης για τους οποίους στόχους δίνουμε μάχη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρέπει η διαφάνεια και η παραπληρωματικότητα, η συμπληρωματικότητα να είναι σημαντικές αρχές, όχι όμως της παραοικονομίας. Το αντίθετο, το, μέσω του blending, του, του μείγματο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρουμε πολύ καλά πόσο χαμηλά επίπεδα διαφάνειας πάγονται όλα αυτά. Ή τους διάβλους που τα δημόσια κονδύλια τα οδηγούν σε ιδιωτικούς, α, ιδιωτικές τσέπες. Πρέπει να το δούμε αυτό. Αν πραγματικά θέλουμε να υπάρξει μόχλευση μέσω των ε, κονδυλίων για τα ιδιωτικά ε, κεφάλαια, Πρέπει αυτό να γίνεται με διαφάνεια και έναν υγιή τρόπο και να δούμε πώς θα επιτευχθεί αυτό πιο αποτελεσματικά. Πέρα από αυτό έχουμε και κάποιες θέσεις που έχουμε και προτείνουμε για παράδειγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μηχανισμούς ρυθμιστικούς, ρύθμισης ώστε να καταπολεμηθεί η αδιαφάνεια και η φοροδιαφυγή και πρέπει να δούμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εργάζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες ότι πολλές φορές τα κονδύλια τους τα οδηγούν αλλού. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το τι γίνεται σε σχέση με τις, ε, ε, τα δημόσια κονδύλια και τις, ε, την δραστηριοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα υποφεληθούν από τέτοιες δράσεις καθώς επίσης βλέπουμε πολύ συχνά από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν γλωσσικοί φραγμοί πολλές φορές ε, όσον αφορά την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλειών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο είναι μεγάλο σφάλμα. Επίσης πρέπει να στοχεύουμε στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς που είναι αναγκαίοι για την ανάπτυξη όπως ο υγειονομικός τομέας, ε, οι παροχές ε, υπηρεσιών στον τομέα της υγείας για παράδειγμα και την παροχή νερού. Εδώ θα πρέπει πρέπει να δούμε τη δυνατότητα αποτελεσματικών ιδιωτικών επενδύσεων. Θέλουμε να αλλάξει και η ευθύνη της εταιρική ε, ευθύνης από πλευράς επιχειρήσεων έναντι ε, ευθυνών έναντι της κοινωνίας. Να δούμε μια άλλη προσπάθεια για την ανάπτυξη ώστε να καθορίζονται σαφέστατα οι αρχές που θα μπορούν να είναι για παράδειγμα οι ε, αρχές της ε, διεθνούς, ε, ε, του διεθνούς θεματολογίου για την ανάπτυξη και να συνεισφέρουμε έτσι με την προσυπογραφή και υλοποίηση αυτών των αρχών και όρων για την ανάπτυξη. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Ρίκε Γκερέρο παρακαλώ, έχει τον λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ακούστηκαν λοιπόν απόψει ε, τις οποίε δεν θα επαναλάβω από τους προλαλήσαντε συναδέλφου Να ευχαριστήσω έτσι και αλλιώ τον κύριο Ντέβα για την προσπάθεια την οποία έκανε. Είναι αλήθεια ότι σε αυτήν την Επιτροπή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία στην διαδικασία την αναπτυξιακή. Ε, νομίζω ότι ο άνθρωπος πίσω από την προσπάθεια αυτή είστε εσείς η πολιτική μου ομάδα και η προσωπική μου θέση λέει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, προκαταλήψεις και κάποιες ιδεολειψίες αλλά ε, υπάρχουν όμως και κάποιες ε, συγκεκριμένοι κανόνες, κριτήρια που θα πρέπει να οδηγούν στην προοπτική της ανάπτυξης κυρίως και όχι τόσο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι καλοδεχούμενη για να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των χωρών που την έχουν ανάγκη. Όμως θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες λύσεις ε, τις οποίες μπορούμε να συμβιβαστούμε. Πρώτον, να υπάρχει μια συμπληρωματική συνεισφορά στην δημόσια παρέμβαση, να μην αντικαθιστά την δημόσια παρέμβαση. Πάρα πολύ συχνά σε ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε ότι κάποιες κυβερνήσεις συντηρητικές προσπαθούν να προσανατολίσουν κάποιες δραστηριότητες παραγωγικού και επιχειρηματικού τύπου ε, ενώ δεν ευνοούν την δημόσια παρέμβαση. Το θέμα δεν είναι να αντικαταστήσουμε το ένα από το άλλο, είναι να το συμπληρώσουμε. Να μην υπάρξει δηλαδή μία απομάκρυνση και μία μείωση της δημόσιας συμμετοχής στην προσπάθεια για την ανάπτυξη. Δεύτερον, η συγκεκριμένη αυτή ιδιωτική δραστηριότητα θα πρέπει να συμμερίζεται τις βασικές αρχές καταπολέμησης της πείνας, της μάχης για την αηφόρο ανάπτυξη, της καταπολέμησης του αποκλεισμού και της προσπάθειας μείωσης των ανισοτήτων. Εφόσον γίνουν σεβαστές επίσης και οι βασικές αρχές της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας και οι βασικές αρχές της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει πράγματι να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που είναι τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει δηλαδή να ζητήσουμε να υπάρξει μια συμμετοχή των πολυεθνικών και των μεγάλων γενικότερα επιχειρήσεων. Τώρα αν θα μιλήσουμε για social accountability, αν θα μιλήσουμε για κοινωνική ευθύνη, το θέμα είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να έχουν σαν στόχο και υποχρέωση να εξυπηρετήσουν τους πολίτες σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα μέρη στις οποίες δραστηριοποιούνται. Το ε, ιδιωτικό κέρδος το οποίο διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να κυριαρχεί εις βάρος της ευθύνης την οποία έχουν οι επιχειρήσεις αυτές σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών. Τέλος, θα πρέπει επίσης να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της ανισότητας και της προστασίας των περισσότερο ε, θα έλεγα ε, ευάλωτων κατηγοριών των πολιτών. Ευχαριστώ να πω και εγώ λίγα λόγια. Συμφωνώ πως είναι σημαντικός ο ιδιωτικός τομέας σε οποιαδήποτε οικονομία σε εμά και αφρικανικές χώρες ε, χρειάζονται σωστές οργανωμένες κοινωνίες και μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε, αλλά νομίζω πως θα πρέπει επίσης ε, να προσέξουμε το, το ρυθμιστικό περιβάλλον, γιατί βεβαίως πράγματι καλό είναι να δίνουμε 32 δισεκατομμύρια για το νερό, αλλά έλεγξα το νούμερο. Οι τράπεζες κόστησαν στον Ηνωμένο Βασίλειο 850 δισεκατομμύρια λίρες για να ξελασπώσουν τις Βρετανικές τράπεζες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ρυθμιστικό περιβάλλον αυστηρό γιατί μιλάμε για διαφθορά και τα λοιπά. Είχαμε και εμείς τα δικά μας σκάνδαλα, Λάιμπορ και τα λοιπά. Και νομίζω πως ε, είναι μέρος αυτό της συζήτησης για τους στόχους της χιλιετίας. Μιλάμε για κοινά προβλήματα σαν κοινό πλανήτη και βεβαίω ε, εδώ πέρα πρέπει να μπαίνει και η συνεισφορά των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ναι, ο ιδιωτικό τομέας βγάζει τα λεφτά του για του ε, μετόχους του, αλλά οι εταιρείε πληρώνουν του φόρου του, λειτουργούν σε μια κοινωνία και πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη. Γιατί διάβασα μια έκθεση για τη ΣΥΠΑ, όπου ε, εργαζόμενοι πλέον είναι τόσο φτωχοί και δεν μπορούν να αγοράσουν τα αγαθά τους για να λειτουργήσει η Αμερικανική αγορά. Υπάρχει λοιπόν αποσύνδεση ε, των μισθών από την οικονομική ανάπτυξη. Και ε, γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γκερέρο. Δεν είναι θέμα ιδεαλισμού, αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα. Εάν δεν αμείβονται σωστά οι άνθρωποι. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε ένα σύστημα δίκαιο με ανταπόδοση στο κράτος ε, και πιο δίκαιη κατανομή για να μπορεί ο κόσμος να αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες. Φερνόμαστε προσεκτικοί στη χώρα μου, το είπε και η Σίλβα Περέιρα για τις ΣΔΙΤ. Γιατί τι γίνεται, το ξέρω, το έχω δει, αγοράζει φτηνά ο ιδιωτικός τομέας, αγοράζει τη γη και μετά τον δανείζει στον δημόσιο τομέα και παγιδεύεται μετά σε αυτές τις συμφωνίες ο δημόσιος τομέας ε, που είναι μακροχρόνιες. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί να μην αφήσουμε να διαλέγουν αυτά τα οποία θέλουν, να διαλέγουν μόνο τα κέρδη δηλαδή και να αποφεύγουν το ρίσκο. Και βεβαίως ε, κάποια πράγματα γίνονται καλύτερα από τον ε, ιδιωτικό τομέα, κάποια άλλα καλύτερα από τον δημόσιο. Και έχουμε δει τι έγινε τα τελευταία δέκα χρόνια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπα κάποια πράγματα κάνει καλύτερα ιδιωτικό τομέα, ε, τηλεφωνία κτλ. Ακούσαμε από τη UNICEF ε, όσοι είχατε έρθει το μεσημέρι το τι γίνεται με την καινοτομία, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και να φροντίσουμε να μην υποκαθιστά τις δημόσιες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Ντέβα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγγνώμη. Να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλετε να παρεύετε πιο πριν. Έχετε κάτι να πείτε. Εσείς κύριε Ντέβα λοιπόν. Είναι ιδιαίτερα αξιόλογο αυτό που είπατε και το σημειώνουμε όπως πρέπει πρόεδρε. Όλα αυτά που σημειώσαμε θα αναλυθούν στη δράση μας ε, ως πρωτοβουλία μια άμεση απάντηση. Αναφέρθηκε ο όρος διάλογος. Ξέρετε έχουμε μια πολιτική, ένα φόρουμ, ένα βήμα για την πολιτική, για την ανάπτυξη. Διαρθρωμένος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και άλλους εμπλεκόμενους που ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει ακόμα διαδραματίσει το ρόλο που πρέπει και έπρεπε. Ξεκινούμε, προσπαθούμε να βρούμε τον αντιπροσωπευτικό αυτό χαρακτήρα αυτού του φόρουμ. Ξεκινήσαμε τον προηγούμενο Οκτώβριο, θα συνεχίσουμε αναφορά είναι στις νεότερες γενναίες και την παιδεία και κατάρτιση. Και αυτό αποτελεί άρρηκτα τμήμα της φιλοσοφίας και των αρχών που μας εμπνέουν. Η δημόσια παρέμβαση στην εξειδίκευση, στην κατάρτιση τόσο χρήσιμος για τον ιδιωτικό τομέα είναι υποχρέωσή μας να αυξηθεί το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό. Συμφωνώ απόλυτα με την παρέμβαση που έγινε για το CSR. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από το CSR πράγματι αυτή η προσπάθεια. Όταν έχουμε στην προσπάθεια αυτή ανθρώπους που μας σχολιάζουν αυτό το θέμα από για παράδειγμα εταιρική ευθύνη κοινωνική εταιρική ευθύνη που πρέπει να διασφαλίζεται από πλευράς των μεριδιούχων και ομολογιούχων Πράγματι πρόκειται εδώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη βάση της πυραμίδας την ίδια. Η δράση υπαριθμών 11 που έχουμε στην ανακοίνωσή μας που απαριθμούμε επαγγελματική κατάρτιση στην δράση 3. Αυτά που είπατε τα βλέπουμε να αντανακλώνται σε αυτά που απαριθμίσαμε ως προτάσεις και θέσαμε στην προσοχή, υποπροσοχή δική σας. Η πράσινη οικονομία θα μας δώσει μία διάβλο. Διαφέρει από την ε, φεά οικονομία την καφέ οικονομία. Θα πρέπει να παράσχει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ όσον αφορά τις επενδύσεις που θα διασφαλίζονται και θα επιτυγχάνονται. Για το άλλο θέμα, προς να αντιμετωπιστούν τα θέματα διαφάνειας και τους άλλους ε, στόχους ε, για το δημόσιο και ευθυγραμμίζοντας ε, τις μικρομεσές, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις μας δεσμεύουν αυτές οι αρχές για αυτές τις δράσεις. Αυτό που ζητούμε και ρωτάμε οι δικές σας δράσεις θα στοχεύουν στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Αν οι δράσεις σας συνεισφέρουν για την υλοποίηση αυτών των στόχων, τότε μπορούν να ληφθούν υπόψη και να συνυπολογιστούν τι γίνεται, δίνουμε λέει κονδύλια σε εταιρείε. Όχι, δεν δίνουμε χρήματα σε εταιρείε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιε καταστάσει όπου πρέπει να λάβουμε αποφάσει. Αν μα ικανοποιεί τα όσα τεκταίνονται ή όχι. Η, η ηλεκτροδότηση στην Ήπεθρο είναι αυτό που θέλω να υπογραμμίσω και να θέσω ε, ενώπιον τη προσοχή σα. Άλλοι λένε η σορευτικότητα και η προσθετικότητα είναι κριτήριο όσον αφορά την ανακοίνωση. Σορευτικότητα και προσθετικότητα τι σημαίνει. Θα παρεμβαίνουμε μόνο αν διασφαλίζεται ότι χωρίς δική μας παρέμβαση μια επένδυση, μια δράση δεν θα υλοποιείται. Και για την ηλεκτροδότηση αυτό πρέπει να το δούμε. Καθώς μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας ιδιωτικός τομέας που να επενδύει για να έχει πρόσβαση ο πληθυσμός της υπαίθρου στην ηλεκτροδότηση. Γιατί, Γιατί υπάρχουν ε, οικονομικοί παράγοντες ε, που παρακολύουν αυτές τις επενδύσεις. Τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε πάνω από 30 χρόνια για να δοθεί ηλεκτρική ενέργεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, έχουμε υποχρέωση να το πετύχουμε νωρίτερα. Δεν θέλουμε μόνο η προσέγγιση ΜΚΟ να, να λειτουργεί, είναι σημαντικές οι ΜΚΟ και μπορούν να συνεχίσουν και πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους. Όμως με ιδιωτικέ επιχειρήσεις θέλουμε να διασφαλίσουμε αυτό το έργο που πρέπει να στεφθεί με επιτυχία με κριτήρια και αρχές για το συντονισμό με τα ιδιωτικά κεφάλαια θα δράσουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. Καταπολέμηση φοροδιαφυγής, περιβάλλον, λογοδοσία, προστασία του περιβάλλοντος, λογοδοσία, την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να διασφαλίζεται. Ολοκληρώνω πρόεδρε. Πολύ συγκινητική ήταν η παρέμβασή σας σε σχέση με τους καταναλωτές και τα δικαιώματά τους και την, την δυνατότητα να δράσουμε ώστε να διασφαλιστούν. Δεν έχω κομμένη και ραμμένη την απάντηση. Είμαστε πολύ προσεκτικοί για την προσέγγιση του ιδιωτικού τομέα και τη δράση του για τους λόγους που προαναφέρατε. Ξέρουμε ότι υπάρχει κίνδυνος καταχρήσεων, υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν κάποιες αντικαταστάσεις ή υποκαταστάσεις που δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν. Διότι σε σχέση με κάποιες δράσεις δεν θέλουμε να σημειώνονται τέτοια γεγονότα. Θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί σε σχέση με την αγορά. Ένα πολύ σημαντικό μέρος των δράσεών μας θα είναι στο ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και για τον πυρήνα των θεμάτων αυτής της ανακοίνωσης. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε σημαντικά αξιόλογα αποτελέσματα καθώς ε, αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε καταφέρει, ας είμαστε ειλικρινοί, το OVA δεν έχει πετύχει να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα και σε σχέση με τις ε, επιστροφές ε, ε, κάνουμε λόγο εδώ για άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις στην Αφρική αλλά πολύ περισσότερα κονδύλια φεύγουν από την Αφρική, δραπετεύουν από την Αφρική παρότι εκείνα τα οποία εισραίουν στην Αφρική. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο ώστε να πάψει η διαρροή κεφαλαίων από την Αφρική. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ζητούμε λοιπόν να δημιουργηθεί ένα ώστε να υπάρξει εταίρος σε αυτό το διαρθρωμένο πλαίσιο ε, με, για τα ιδιωτικά κεφάλαια. Και ζητούμε λοιπόν προς αυτή την πορεία να πορευτούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίρτς Ντέβα. Νομίζω όταν ακούω να ομιλεί εκπρόσωπος της Επιτροπής με τέτοιο πάθος νιώθω πράγματι ενθουσιασμένος. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για όσα τα ενδιαφέροντα είπατε. Για... Ο Ενρίκο είπε ότι προσπάθησα εγώ να βάλω ε, εδώ και πολύ καιρό τον ιδιωτικό τομέα στον χώρο της ανάπτυξης και θα του απαντήσω γι' αυτό. Εγώ έκανα κάποιες απλές πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προϋπολογισμός της φέτος είναι περίπου 145 εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια, ένα ποσοστό δηλαδή, το οποίο είναι 1,05 περίπου ε, του συνόλου δίδεται για την ανάπτυξη. Εμείς επανειλημμένα έχουμε εκφράσει το αίτημα Ε, ότι πρέπει να φτάσουν οι χώρες αυτές το 0,7 του δικού του ΑΕΠ στο, ε, στην ανάπτυξη. Αν το κάνουμε αυτό θα φτάσουμε 140 δις. Το 140 δις είναι 1,1 και 120 είναι το 0,7 περίπου. Το σύνολο λοιπόν στο οποίο αναφερόμαστε τώρα ε, φτάνει περίπου τα 120 δις γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο δισεκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο που ζουν με ένα με δύο δολάρια την ημέρα. Σε ένα πραγματικά παράδεκτο επίπεδο φτώχειας. Δεν χρειάζεται ε, επιστήμη ιδιαίτερη για να διαιρέσει τα 100 τόσα δις από τη μία με τα δύο από την άλλη για να δει ότι μιλάμε για 65 ευρώ το χρόνο στον καθένα. Λοιπόν, η Επιτροπή μας, η κοινότητα, η αναπτυξιακή, όλες οι ΜΚΟ, εμείς τι συζητάμε, συζητάμε το να δώσουμε 65 δολάρια το χρόνο σε αυτούς τους δύο δις φτωχούς που ζουν με ένα με δύο δολάρια την ημέρα. Ένα ευρώ δηλαδή τη βδομάδα τους δίνουμε ουσιαστικά. Και κάνοντας το αυτό, εμείς στην ουσία λέμε ότι θα καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Κάνουμε χιλιάδες συναντήσεις ε, για την σύνολη ανάπτυξη, θέματα εν πάση περιπτώσει συνδυασμού των πόρων. Έχουμε τρομερές δαπάνες γύρω από αυτά για να δώσουμε στους φτωχούς αυτούς, τους πολύ φτωχούς, ένα ευρώ τη βδομάδα. Ε, έτσι δεν θα αντιμετωπίσουμε ε, με 65 ευρώ το χρόνο τη φτώχεια, είναι παράλογο. Είναι χαζότο να το πιστεύει κανείς. Εμείς χρειαζόμαστε κάτι το διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τα κράτη-μέλη δεν θα δώσουν περισσότερα χρήματα, δεν θα φτάσουν το 7%, ίσα ίσα φεύγουν από το 0,7% και με αυτά τα 120 δις ε, που δεν είναι ήδη ε, πραγματικότητα. Ούτε καν 65 δηλαδή ευρώ ε, τον χρόνο. Ακόμα και λιγότερο από αυτά. Όταν κάνουμε ό,τι κάνουμε αυτό είναι όλο και όλο. Γι' αυτό λοιπόν προσπάθησα να δω με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που ζουν ακριβώς με στη ζητιανιά ε, σε απαράδεκτες καταστάσεις εδώ και πάρα πολλές γενιές, χωρίς ελπίδα. Είχαμε λοιπόν μια πολύ θετική συζήτηση και συγκινήθηκα από κάποια από αυτά τα οποία ακούστηκαν. Αυτό που είπε η Λάιλα για τη φοροαποφυγή είναι πάρα πολύ σωστό. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους χώρους τους οποίους είναι εγκατεστημένες και να μην πληρώνουν φόρους γιατί έχουν ε, υπεράκτιες έδρες των επιχειρήσεων ευρωπαϊκές, αμερικάνικες και θα πρέπει να μην συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει να πληρώσουν τους φόρους στις τοπικές αρχές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης και το θέμα της πρόσβασης στην πίστοση, όπως είπε ο Σίλβα Περέιρα. Θα πρέπει να εξετάσουμε θέματα σύνολης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αυτό που είπατε για την κατάρτιση και τη βιοτεχνία. Μετά τον πόλεμο στη Σρι Λάνκα, η Σρι Λάνκα έχει ρυθμό ανάπτυξης 14% και στο βορρά που ήταν ο πόλεμος αναπτύσσεται με 25%. Αν πάτε στο Σρι Λάνκα σήμερα θα δείτε παντού γερανούς, οικοδομούν κτλ. Ζητώ από αυτούς λοιπόν, έχετε αρκετούς ξυλουργούς, και μου λένε όχι βέβαια, δεν έχουμε, εμείς τους εκπαιδεύουμε με ταχύτητα. Φτιάχνουμε τεχνικά σχολεία για ξυλουργούς, για ηλεκτρολόγους κτλ. Λοιπόν, και είπα στις μεγάλες επιχειρήσεις, εσείς τους βοηθάτε να φτάσουν στα επίπεδα τα οποία χρειάζεται ή απλά τους μαθαίνετε να τα βολεύουν απλά τα πράγματα λένε ότι αν φέρουμε τις διεθνείς επιχειρήσεις για να εκπαιδεύσουν ε, τα παιδιά σε αυτές τις μικρές σχολές, ε, τότε στην ουσία θα έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε. Να δώσουμε τη σωστή κατάρτιση μέσω του ιδιωτικού τομέα. Είμαι ευγνώμων στην κυρία Χάουταλα για τα θετικά της σχόλια και θα συνεργαστώ μαζί της. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Νορμπέρ για αυτά τα οποία είπε για τις σωστές επιχειρήσεις και τις νέες γενιές και πώς μπορεί να εκπαιδευτούν σωστά οι νέες γενιές. Και επίσης είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και από αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως για τον εξηλεκτρισμό της Υπέθρου. Εμείς περιμέναμε 50 χρόνια για να έρθει το ρεύμα από 300 χιλιόμετρα στην Αφρική. Εγώ είχα πάει στον Μπραζαβίλ εδώ και λίγο καιρό και η περιοχή είναι πραγματικά μικρούς καταράχτες. Και είπα στους υπουργούς, πού είναι τα μήνυ υδραυλικά σας έργα και μου είπε τι είναι αυτά, γιατί συζητάς. Εγώ έβλεπα, έβλεπα ε, τα τοπικά χωριά να αγοράζουν τους μικρούς καταράχτες ε, και να φτιάχνουν ένα μήλο υδρόμηλο παραγωγής ρεύματος για να εξηλεκτρήσουν το χωριό τους, αλλά δεν το σκέφτονται αυτό. Αυτό είναι που είπε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Αν δώσουμε μικροπιστώσει στο χωριό αυτό για να αγοράσει μια μικρή εγκατάσταση, τότε πράγματι ε, μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες θα προχωρήσουν. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλά που είναι εφικτά σήμερα να γίνουν. Η μεταφορά είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα σε σχέση με τη σύνταξη αυτής της έκθεσης προσβλέπω στις τροπολογίες είναι υποεξέλιξη όμως εξέλιξη η φάση σύνταξης δεν μπορεί να είναι σε μια δεδομένη στιγμή όλα να αναφέρονται και να είναι πλήρης μια ε, έκθεση πρέπει λοιπόν μακροπρόθεσμα να προσεγγίσουμε το εγχείρημα να υπάρξει πρόσβαση λοιπόν σε κεφάλαια και χρηματοδότηση πρόσβαση στα χρήματα είναι κάτι παράλογο και τρελό να νομίζει κανείς ότι με 65 ευρώ ετήσια ή 1 ευρώ ανά εβδομάδα θα λύνει προβλήματα, θα λύσει, θα λυθούν προβλήματα στην Αφρική. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πράγματι διαβάσαμε την έκθεση αυτή και τις άλλες δύο εκθέσεις για τη φορολογία και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Πρέπει να ορίσουμε ξεκάθαρα ποια έκθεση θα κάνει το τι αλλιώς θα καλύπτουν όλες τα πάντα. Πρέπει να τα μοιράσουμε λοιπόν. Ε, θα βρει η γραμματεία έναν τρόπο να μοιράσει τα θέματα αυτά και όλο το πακέτο νομίζω είναι συνεκτικό ε, για να είναι συνεκτικό με τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε λοιπόν και όπως είπες υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία αλλά έχουμε αυτές τις τρεις εκθέσεις. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Υπάρχει συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια για το Νότιο Σουδάν. Θα υιοθετηθεί ψήφισμα αύριο το βράδυ. 17 Νοεμβρίου, 5 η ώρα, ο κύριος Λιανίδης θα έρθει να μας πει τι είδε στη Δυτική Αφρική για την έμπολα. 24 Νοεμβρίου, ειδική ακρόαση στο Στρασβούργο με τον ε, δόκτωρα Μακου, το γιατρό Μακουέγγι που πήρε το βραβείο Ζαχάροφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύσκολη μέρα, αλλά νομίζω ήταν παραγωγικές συζητήσεις. Ευχαριστώ τους ερμηνείς. Τελειώσαμε και πέντε λεπτά νωρίτερα. Οπότε νομίζω έτσι σας εξοφλώ για τις υπερβάσεις που είχαμε κάνει. Ευχαριστώ.